Dear Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλες οι παρούσες και όλοι οι παρόντες, business as usual. Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ενέργειας. Μη λησμονείτε ότι μεταδιδόμαστε και από το διαδίκτυο διαρκώς. Ας αρχίσουμε λοιπόν αμέσως γιατί έχουμε σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη μας σήμερα. Την ε, ημερήσια διάταξη θα τη βρείτε στους φακέλους σας. Με ακούτε ή δεν με παρακολουθείτε καθόλου. Ρωτάω ο πρόεδρος Μπούσικ. Δεν μου αρέσει να κτυπώ την σφύρα, αλλά χρειάζεται κάποια ησυχία διότι είναι αδύνατον να με ακούσετε αν δεν χρησιμοποιήσω το εργαλείο τούτο. Εννοεί τη σφύρα. Όπω έλεγα λοιπόν, η μερισία διάταξη περιλαμβάνεται στου φακέλου των Ευρωβουλευτών. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, μπορούμε να την εγκρίνουμε χωρί περαιτέρω αλλαγέ. Επιθυμείτε να πείτε κάτι για την ημερησία διάταξη? Όχι, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν εγκρίνεται την ημερησία διάταξη. Δεύτερο θέμα τώρα, ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχουμε τέτοιες. Διότι την προηγουμένη εβδομάδα κάναμε τη συνεδρίασή μας και έχετε λάβει όλα τα σχετικά. Έτσι λοιπόν έρχομαι στο 3 που το επιγράφεται δημιουργία Ενεργειακής Ενώσεως. Καλώς ήλθατε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Μάρος Σεύκοβιτς, Αντιπρόεδρος για θέματα Ενεργειακής Ένωσης. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Μάρος, σας έχουμε υποδεχτεί κατ' επανάληψη εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία. Το ίδιο τη φορά, ωστόσο, με νέο χαρτοφυλάκιο ευθυνών δικό σας. Την προηγουμένη φορά ήταν η αρμοδιότητά σας για τη διαθεσμική συνεργασία. Τώρα είστε αντιπρόεδρος, αντιπρόεδρος σας δηλαδή και στην προηγούμενη θητεία βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα όμως έχουμε την Ενεργειακή Ένωση, βασική σας ε, ευθύνη και δική μας. Και είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε μια σοβαρή και σε βάθος συζήτηση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα που είναι από τις πιο κέρυες ιδέες για τα επόμενα πέντε χρόνια του Ευρωκοινοβουλίου, βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου των Υπουργών. Για να μπορέσει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, έχουμε προβλέψει δύο ώρες για όλη τη συζήτηση. Λογαριάζω δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και μετά θα προχωρήσουμε σε συζήτηση. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος ε, ε, Σεύκοβιτς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα-πρώτα ομολογώ ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την παρουσία σας, από το ενδιαφέρον σας, από το μεγάλο αριθμό των παρουσών και παρόντων που επιθυμείτε να συζητήσουμε την Ενεργειακή Ένωση. Γι' αυτό και ευχαριστώ ιδιαίτερος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα την Επιτροπή Ενέργειας που οργάνωσε την έκτακτη αυτή συνεδρίασή σας, διότι το σχέδιο της Ενεργειακής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες και το ίδιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της ε, Επιτροπής Juncker και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα εν συντομία λίγες από τις ιδέες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε τώρα και πιο σημαντικό βέβαια οι δικές σας προτάσεις με ενδιαφέρουν γιατί οι προτάσεις και οι ιδέες ξεπηδούν μέσα από τη συζήτηση και γνωρίζω ότι πολλοί από εσά είστε σε θέματα ενέργεια. Γι' αυτό επιθυμώ να τονίσω ότι έχω προσέλθει εδώ και για να ακούσω, να σημειώσω τις προτεραιότητες, τις ανησυχίες και τις ιδέες σας. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσά συντάσσετε γραπτές θέσεις για την Ενεργειακή Ένωση. Άλλοι και άλλες από εσά θα έλθουν σε προσωπική επαφή μαζί μου για να συζητήσουμε και ήθελα να σας πω ότι εγώ προσωπικά είμαι πανέτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας. Η σημερινή μας συνάντηση είναι και πολύ επίκαιρη, διότι μόλις προ δύο εβδομάδων, μάλλον σε λίγες εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες, συγγνώμη, θα δώσουμε τελική μορφή στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θα σας τα πω και μετά από τη σύντομη εισαγωγή μας. Το χρονοδιάγραμμά μας ελπίζω ότι θα υποβληθεί η πρόταση και θα εγκριθεί από το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων 5 τέλη Φεβρουαρίου. Θα συζητήσουμε τότε με τον πρόεδρο Μπούσεκ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε πρώτους εσάς για το σχέδιο της Ενεργειακής Ένωσης, να φτιάξουμε δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η συζήτηση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Επιτροπής, ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αξιότιμες φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέλαβε τώρα, ανέλαβε λέγοντας ότι θα φανεί μεγάλη στα μεγάλα πράγματα για τα θέματα και τις πολιτικές εκείνες δηλαδή που έχουν βαθιές επιπτώσεις στις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε εν τέλει η θέρμανση των σπιτιών να είναι ευθυνή, να μπορεί να την πληρώσει ο πολίτης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε μα, οι επιχειρήσει μα και οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να μπορούν να αγοράζουν την ενέργειά του σε ανταγωνιστικέ τιμέ και να αποδειχτεί ότι αυτέ είναι οι κινητήριε δυνάμει για την ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η μεγαλοφία του και του Πόρτο να μπορέσει να κάνει πρόοδο, να προχωρήσει επιστημονικά εδώ στην Ευρώπη, αντί να χρειάζεται να πάει στις ΗΠΑ ή στην Κίνα για να το πετύχει αυτό. Και θέλουμε τελικά να εξασφαλίσουμε ότι τα δικά μου παιδιά στην Πρατισλάβα, τα δικά μας παιδιά σε όλη την Ευρώπη, απανταχού της Ευρώπης και στο τελευταίο χωριό της Ευρώπης, ότι δεν θα χρειαστεί τα παιδιά αυτά και τα εγγόνια μα να πληρώσουν το τίμημα των περιβαλλοντικών σφαλμάτων που έκαναν οι προηγούμενε γενιές. Ίσως οι στόχοι αυτοί να σα φανούν φιλόδοξοι. Όμως μπορούμε να του επιτύχουμε και το πολιτικό κλίμα υπάρχει για να βάλει μπρο επιτέλου η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ενεργειακή Ένωση. Η γεωπολιτική κατάσταση στα ανατολικά μα σύνορα, παρόλο που είναι ιδιαίτερα ατυχή, έχει βάλει ωστόσο την ενέργεια πολύ ψηλά στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για το πλαίσιο του 2030, για το κλίμα και την ενέργεια. Και για το Παρίσι διαγράφονται καλές οι προοπτικές, αφού και άλλοι ηγέτες ανά τον κόσμο θα συνεργαστούν. Έχουμε και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα δώσει όθηση για να υπάρξει μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση στραμμένη προς τα εμπρός. Το σχέδιο επενδύσεων Juncker, που είναι σχεδιασμένο για να ξεκλειδώσει εντό εισαγωγικών τα χρηματοδοτικά μέσα για τον τομέα της ενέργειας, να φτάσει δηλαδή στην κρίσιμη κίνη μάζα πολιτικής βούλησης που θα επιτρέψει να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και επομένως να επέλθει μια σοβαρή διαφορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα καταφέρουμε. Τώρα έχει έρθει η στιγμή να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή. Κυρίε και κύριοι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια, πράγματι έχουμε κάνει πρόοδο, όμως πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Και για να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι οι τρέχουσες ενεργειακές πολιτικές μας δεν είναι βιώσιμες, με κανένα τρόπο, με καμία έννοια. Οι τιμές του πετρελαίου είναι ακατάστατες εντελώς και προκαλούν κερδοσκοπικές τάσεις βραχυπρόθεσμα και αβεβαιότητα μακροπρόθεσμα. Το γεγονό ότι την περισσότερη ενέργεια την εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα από χώρε οι οποίε χρησιμοποιούν την ενέργεια ω πολιτικό όπλο, μα θέτει διαρκώ ενώπιον του κινδύνου των διακοπών παροχή. Βλέπετε και στον πίνακα, στο γράφημα που σας προβάλλουμε στην οθόνη, πόσο πολύ εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, πόσο πολύ εξαρτώμεθα από τρίτες χώρες για την προμήθεια ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 90% του πετρελαίου μας, 66% του αερίου μας, 42% ε, στερεών καυσίμων και 6 χώρες μέλη εξαρτώνται 100% από το φυσικό αέριο που εισάγουν από τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν οριοθετεί γεωπολιτικά το τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την ανεξαρτησία μας την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας, να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες ενέργειες που αυτές είναι οι γηγενεί, εδώ οι θαγενείς μας ενέργειες. Πρέπει να είμαστε επίσης ειλικρινείς και να πούμε ότι τα ενεργειακά μας συστήματα είναι κατακαιρματισμένα σε 28 ξεχωριστές μονάδες και ορισμένα τμήματα της υπήρου μας πόρο απέχουν από το να είναι ενταγμένα στα ενεργειακά συστήματα. Αν δείτε τούτην εδώ τη διαφάνεια τώρα, θα δείτε τις διαφορετικές πολιτικές που ασκούν οι διάφορες χώρες ή και οι διάφορες περιφέρειες. Στις προτάσεις που κάνουν για ε, τους μηχανισμούς ικανοτήτων, capacity mechanisms δηλαδή. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να φτάσουμε στο κατάλληλο επίπεδο των μηχανισμών αυτών, αλλά Χρειάζεται να φτιάξουμε τέτοιου capacity mechanisms απανταχού της Ευρώπης σε κάθε χώρα. Χρειάζεται να πληρώσουμε το υψηλό αυτό κόστος για τη δημιουργία των μηχανισμών αυτών ή να αναζητήσουμε καλύτερα κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η Ευρώπη στην περίπτωση αυτή, περισσότερη Ευρώπη είναι η λύση. Δέστε τα ε, συστήματα ενίσχυση των ανανεώσιμων ενεργειών πόσο μας έχουν κοστίσει. Και όμως όλοι έχουν κατευθυνθεί προ εθνικά συστήματα. Παρακολουθώ το τι λένε τα διάφορα think tank και διαβάζω διάφορες μελέτες και ένα από τα πράγματα που είναι πραγματικά απίστευτο όταν αρχίσαμε με την υποστήριξη των ανανεώσιμων ενεργειών από την αρχή δηλαδή στο πανευρωπαϊκό επίπεδο αν τα είχαμε κάνει αυτά πανευρωπαϊκά, θα είχαμε εξοικονομήσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα χρειάζεται να κάνουμε πιο, αποτελεσματική, ε, πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό στο μέλλον. Άλλο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι ενώ πολλοί εξημών και μετά από τη συνάντησή μας εδώ θα γυρίσουμε στα ζεστά μας σπίτια ή ξενοδοχεία, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών νοικοκυριών που δεν μπορούν να θερμανθούν, διότι οι ενικοί τους δεν μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια για να ζεσταθούν. 10% των ε, νοικοκυριών μας είναι φτωχά τόσο που δεν μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια που χρειάζονται. Θέλουμε λοιπόν να λυθεί και το πρόβλημα αυτό. Βεβαίως δεν είναι μονάχα οι καταναλωτές, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πληρώνουν τιμές φυσικού αερίου τριπλάσιες από τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Τεράστιο βάρος αυτό στους ώμους της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας. Και όταν μιλούμε για την βιομηχανία μας, από τις 10 top εταιρείε ηλιακής ενέργειας, καμία δεν είναι ευρωπαϊκή. Επίσης καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια στην Ευρώπη και δεν έχουμε φτιάξει ακόμα την οικονομία και κοινωνία εκείνη που θα καταναλώνουν λίγο πετρέλαιο, θα εκλείουν λίγα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Όπως, όπως σας ανέπτυξα και στη διάρκεια της ακροάσεώς μου, η Ενεργειακή Ένωση που οραματιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που σας περιέγραψα, θεωρώ ότι έχει πέντε διαστάσεις που είναι αλληλοσυμπληρούμενες και συνδεδεμένες. Και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα προτείνουμε και συγκεκριμένες δράσεις για κάθε μια από τις διαστάσεις αυτές. Λοιπόν, η πρώτη είναι η ανάγκη αύξησης της ασφάλειας προμήθειας ενέργειας βασισμένη στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη. Είμαστε η μεγαλύτερη εισαγωγή ενέργειας στον κόσμο. Κάθε χρόνο δαπανούμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αγωγές ενέργειας. Άρα χρειάζεται μείωση για να γίνει, της εξάρτησης αυτής. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας και καλύτερη χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Θυμηθείτε το πρόσφατο αυτό θρύλο του ε, αγωγού South Stream και ας μας γίνει μάθημα. Να βάλουμε περισσότερη διαφάνειας, της αδιαφανής συμβάσεις για το φυσικό αέριο και μαζί με την κυρία Μογκερίνη ας σχεδιάσουμε μια συνεπή ενεργειακή διπλωματία στην, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε και ο μεγαλύτερος πελάτης του κόσμου τελικά. Χρειάζεται λοιπόν να μας αντιμετωπίσουν και με, με τον απαραίτητο σεβασμό. Η δεύτερη πρότασή μας θα είναι να δημιουργήσουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας που να είναι έντονα ανταγωνιστική. Γνωρίζετε ότι έχουν βήματα αλλά μένουν πολλά ακόμα. Χρειαζόμαστε μια αγορά μέσα στην οποία η ενέργεια να ρέει ελεύθερα. Με τις καλύτερες ενεργειακές τιμές, με σεβασμό κοινωνιακών και ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Και επομένως πρέπει να πέσουν οι φραγμοί μεταξύ των χωρών μελών. Ως πρώτο βήμα θα δημιουργήσουμε μια στενότερη περιφερειακή συνεργασία μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στη βάση συζητήσεων που διεξήγαγα τελευταία με δημάρχους και με τοπικές εταιρείες ενέργειας είμαι πεισμένος ότι μπορούμε να πετύχουμε την Ενεργειακή Ένωση μόνο με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών παραγόντων και των πόλεων, ευφυών πόλεων. Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις που θα προτείνουμε. Τρίτη σημαντική διάσταση που επιθυμώ να σας θέσω υπόψη είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Όσοι γνωρίζουμε, η πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν χρησιμοποιούμε. Λιγότερη ενέργεια σημαίνει και λιγότερη ρήπανση και διατήρηση των ενεργειακών πηγών μας. Η βελτίωση λοιπόν της ενεργειακής αποδοτικότητας θα βελτιώσει και την ασφάλεια προμήθειας και τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα δηλαδή και την αηφορία. Πάλι εδώ οι καταναλωτές θα βρίσκονται στο επίκεντρο γιατί θα ωφεληθούν από την βελτίωση της αγοράς και από την αυξημένη αποδοτικότητα της ενέργειας. Σε μια πρόσφατη συνάντηση μου είπαν ότι 90% των οικειών μας μου είπαν ότι είναι energy inefficient, δηλαδή κατασπαταλά την ενέργεια. Και μετά, σε άλλη συνάντηση, ιδιώτε επενδυτέ που μου είπαν ότι οι επενδύσει του φτάνουν τα 9-3 εκατομμύρια ευρώ, είναι, πολύ, είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε επενδύσει στην οικονομικότερη χρήση τη ενέργεια, στην αποδοτικότερη χρήση τη ενέργεια. Αυτό χρειάζεται να γίνει. Έτσι επιθυμούν να συνεργαστούν σε αυτό και οι τοπικοί δήμαρχοι, οι τοπικοί φορείς, να μην φοβούνται να αρχίσουν την προσπάθεια αυτή. 40% της ενέργειας που καταναλώνουμε πηγαίνει στη θέρμανση ή στην ψήξη. Ασφαλώς μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα στο μέλλον. Τέταρτη σημαντική διάσταση είναι η ανάγκη μείωσης της έκκλησης αερίων θερμακηπίου από τις οικονομίες μας, από τη βιομηχανία μας. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς το Παρίσι. Και αυτός ο δρόμος περνάει από την Ενεργειακή Ένωση. Τον Οκτώβριο είχαμε συμφωνήσει να μειώσουμε κατά 40% τις εκπομπές των καυσαερίων. Στη Λίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκε και είπατε εκπρόσωπος κυρία Μογκερίνη μαζί με τον Επίτροπο Αρία Κανιέτε και εμένα τον ίδιο θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνεργασία, αυτή η ενία φωνή στη διπλωματία του κλίματος θα είναι καθαρή και δυνατή. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Παρίσι να είναι επιτυχία. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη τα χρειάζεται αυτά, είναι ο ίδιος ο πλανήτης. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και στο σπίτι και ενθαρρύνω όλα τα μέρη να προχωρήσουν σε καλή και φιλόδοξη συμφωνία για, την, ε, για το αποθεματικό σταθερότητα της αγοράς και ιδίως για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των αερίων του θερμοκηπίου. Και πρέπει να κάνουμε βεβαίω και σημαντική προσπάθεια στι ανανεώσιμε ενέργειε. Όπω είπε ο πρόεδρο Γιούνκερ, η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα παγκοσμίω για τι ανανεώσιμε ενέργειε. Πρέπει να μειώσουμε και τι εκκλήσει καυσαερίων του τομέα των μεταφορών. Τελευταία, πολύ σημαντική πάλι διάσταση, πώ μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τι ανανεώσιμε ενέργειε με επενδύσει στην έρευνα και στην καινοτομία. Γιατί εκεί είναι κέρια η έρευνα και η καινοτομία. Όχι μόνο για εναλλακτικέ ενέργειες, αλλά και για να μειωθεί η κατανάλωση των παραδοσιακών ενεργειών. Γιατί έτσι θα αυξηθεί και η ανάπτυξη και η απασχόληση. Γνωρίζω ότι γι' αυτό και για σας είναι σημαντική προτεραιότητα και γνωρίζω ότι θα το συζητήσετε μάλιστα και σήμερα το θέμα αυτό, αμέσως μετά από τη δική μας συζήτηση. Αυτές οι πέντε διαστάσεις απηχούν μια συνολική προσέγγιση μέσα από πολλούς τομείς πολιτικής, από τις μεταφορές, τον ανταγωνισμό, τη γεωργία μέχρι τη βιομηχανική πολιτική. Μέσα στο περιορισμένο χρόνο που έχω δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις πτυχές, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχετε κατανοήσει ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας. Δική μου προσωπική ευθύνη θα είναι να διασφαλίσω ότι αυτές οι διαστάσεις που σας εξήγησα και οι τομείς πολιτικής που τους αναλογούν θα λειτουργήσουν σε αρμονία και με συνεργασία όλων των ε, φορέων γύρω από ένα τραπέζι. Η, η Ενεργειακή Ένωση χρειάζεται και ένα στέρεο και αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης. Διάβασα την επιστολή που στείλατε ορισμένοι από εσά στον πρόεδρο Γιούνκερ, στον κύριο Κανιέτε και σε μένα. Συμφωνώ ότι οι ανησυχίε σα είναι ορθέ, ότι το Κοινοβούλιο ως ένα από τους νομοθέτες έχει κέριο ρόλο να παίξει για να υλοποιήσει την Ενεργειακή Ένωση. Γι' αυτό, σε ένα μήνα περίπου που το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων θα εγκρίνει τις προτάσεις μας, θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου επιτρόπους να προσέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας εξηγήσουν, να αναπτύξουν τις προτάσεις μας. Αυτό θα το πράξω γιατί λογαριάζω και με την υποστήριξή σας. Γιατί αυτή η βαθιά αλλαγή, αυτή η βαθιά μεταρρύθμιση μπορεί να επιτύχει μόνο εάν έχουμε και τη σταθερή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ολοκληρώσω εδώ και πολύ ευχαρίστω να απαντήσω στι ερωτήσει των Ευρωβουλευτών σα. Σα ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Επίτροπε ε, και για την ενθουσιασμό και την ενεργητικότητα με την οποία παρουσιάσατε τα θέματα αυτά καθώς και για τα θεσμικά σας επιτεύγματα. Ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ μας και πόσο σημαντικό είναι που μπορείτε να παρουσιάσετε στους βουλευτές τις ιδέες και τις προτάσεις σας για την Ενεργειακή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ας ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο τους συντονιστές μας. Εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος ε, Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σεύκοβιτς για αυτή την επισκόπηση για το τι επεξεργάζεστε. Όπως ξέρετε η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή Μάζει μια ιδέα πρωτοβουλία ε, έκθεση, συντάσσει μια ιδέα πρωτοβουλία έκθεση που σημαντικό θα είναι να τη λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα της Ενεργειακής Ένωσης. Έχω μια ερώτηση ως προς τα δύο πρώτα σημεία, την εσωτερική αγορά και την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Πριν από δύο εβδομάδε, αν έχω καταλάβει καλά, ήσασταν στη Μόσχα και ο κύριο Σομίλερ ήρθε και σα είπε από το πουθενά ότι φίλε μου, Αρχίστε τον τουρκικό αγωγό τώρα και αρχίστε να τον χτίζετε γιατί σε κανένα δυο χρόνια δεν θα περάσει τίποτε από αέριο από την Ουκρανία. Μια πολύ επικοδομητική σχέση για την ε, προσέγγιση μάλλον για την εταιρική μας σχέση. Αλλά αυτό είναι ο εταίρος που έχουμε απέναντί μας και αυτές τις προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το απρόβλεπτο ουσιαστικά. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει είναι κατακαιρματισμένη η αγορά μας. Όμως, αν μιλάμε για τον εξανατολάς ε, εταίρο μας ε, με έναν εφημισμό, ουσιαστικά εννοούμε τη Ρωσία. Τα περισσότερα κατημέλη αυτή τη στιγμή έχουν ένα διμερή διάλογο με το Ρώσο προμηθευτή. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία με την χώρα Α, μετά είναι διαφορετική με τη χώρα Β, με τη χώρα Γ και ούτω καθεξής. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μαθαίνετε εκ των υστέρων ε, το τι συμφωνίες έχουν ε, γίνει και να κοιτάζετε αν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να έχουμε μια ενωμένη φωνή με την αγορά των 500 εκατομμυρίων για να έχουμε καλύτερη συμφωνία από τη ρωσική πλευρά. Και αν ναι, πώς μπορούν αυτές οι συμφωνίες που τις έχουν σχεδιάσει ιδιωτικέ εταιρείε σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις να οδηγήσουν σε μια άλλη συνδυασμένη προσπάθεια. Γιατί οι ιδιώτες ενδεχομένως να μην θέλουν να μαθευτούν και τα ε, στοιχεία των εταιρεών τους. Εάν λοιπόν ενωθούν οι προσπάθειές μας, όλα θα βελτιωθούν και θα έχουμε ενδεχομένως σημαντικούς όγκους ε, που θα μπορούν να εισαχθούν από την Ανατολή. Τι προτείνετε λοιπόν να μπορούσαμε να κάνουμε, τι προτείνετε να κάνουμε με κάποιον τόσο απρόβλεπτο όπως ο κύριος Μίλλερ. Ευχαριστούμε εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών, ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά μια που έχω την ευκαιρία. Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω Πότε έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό να προχωρήσει στην ανθεώρηση οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την οδηγία για, τις ε, ενεργειακή, για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια. Ήθελα να μου πείτε εάν η νέα πρόταση θα λάβει υπόψη την κατάσταση των ευάλωτων καταναλωτών, των πλέον φτωχών από ενεργειακή πλευρά. Σημειώνω το γεγονό ότι και εσεί και ο κ. Γιούγκερ είπατε ότι χρειαζόμαστε την Ενεργειακή Ένωση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση με σκοπό τη βιώσιμη οικονομία. Έω το 2020 υπάρχουν εκτιμήσει ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα θα είναι ένα σημαντικότατο τμήμα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε, εάν ο στόχο του 20% που έχουμε ήδη ε, θέσει για, τους, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, πώ θα επιτευχθεί, πώ ε, εντάξει εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμά σας. Και έπειτα, εφόσον όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και μάλιστα στην ευρωπαϊκή επικράτεια, εντάξει, αλλά η βιομηχανία που καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντος. Η βιομηχανία αυτή πρέπει να έχει ένα σταθερό πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει, να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ε, ιδιαιτέρως εκτός. Ε, πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, ιδίω επειδή η τιμή της ενέργειας επηρεάζει, επηρεάζει τις οικονομικές δραστηριότητες. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε οι τιμές να είναι κάπως πιο προβλέψιμες στο μέλλον. Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα επιδοτούν ή δεν θα επιδοτούν τις διάφορες μορφές ενέργειας, ιδίω τι ανανεώσιμες. Με αφορμή λοιπόν τα όσα είπατε, να δώσω παράδειγμα την Ρουμανία. Ε, έχουμε ήδη αιωλική παραγωγή αιωλική ενέργειας στη χώρα μας, αλλά πωλείται 10 ή 15% χαμηλότερα από την τιμή της ενέργειας στην αγορά. Διότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην παραγωγή ακριβώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής ε, εξ ονόματος ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ο κ. Γκρομπαλτσίκ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις οι οποίες δείχνουν σαφώς το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον ε, με βάση την Ενεργειακή Ένωση. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι πάρα πολύ απλή. Το γνωρίζουμε αυτό γιατί μιλούσαμε εδώ και καιρό και δεν είναι τίποτα το καινούριο. Θέσατε σημαντικά ζητήματα όπως το θέμα των ανατολικών προμηθευτών. Τι θα γίνει αν σταματήσει η προμήθεια Ενέργεια στην Ευρώπη. Ποια είναι τα εναλλακτικά σενάρια. Έχουμε προετοιμαστεί για εναλλακτικές ε, προμήθειες. Έχετε αξιολογήσει το κόστος. Επίσης, δεν αναφέρατε καθόλου τις ανανεώσιμες. Και όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής πρόκειται για την πιο ακριβή πηγή ενέργειας. Οπότε πώς θα διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών. Και δεν θέσατε βεβαίως το θέμα των πηγών που χρησιμοποιούνται ήδη στην Ευρώπη. Το θέμα λοιπόν μιας ε, οικονομίας χαμηλού άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις παραδοσιακές πηγές. Άνθρακα, αέριο, σχιστολιθικό αέριο. Τι έχετε να πείτε για αυτά τα ζητήματα. Για το θέμα πανευρωπαϊκών τώρα διασυνδέσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι προτείνει η Κομισιόν όσον αφορά την χρηματοδότηση τέτοιων ε, διασυνδέσεων. Έχετε σκεφτεί το θέμα χρηματοδότησης ε, ε, τέτοιων πανευρωπαϊκών διασυνδέσεων που θα μειώσουν τους ενεργειακούς κινδύνους και η Κομισιόν έχει προετοιμάσει τα οικονομικά δεδομένα γιατί είναι σημαντικό και αυτό για εμάς. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Πέτερσεν εξ ονόματος της ΑΛΔΕ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό αυτό το οποίο αναλαμβάνετε να κάνετε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία αφορά την ε, διακυβέρνηση και άλλη τη χρηματοδότηση. Γιατί για να λειτουργήσει το σχέδιο αυτό χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο θα αφορά και την επιβολή της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας. Ε, το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής όλη αυτή η νομοθεσία η οποία βεβαίως πρέπει και να εφαρμοστεί πώς έπεται ε, να επιδρά στην ε, διαδικασία ε, λήψης αποφάσεων το δημοκρατικά ερετό κοινοβούλιο για την εφαρμογή όλης αυτής της νομοθεσίας. Και βεβαίως τι σκοπεύετε να κάνετε, θα υπάρξει κάποια συναπόφαση του Κοινοβουλίου, πώς το βλέπετε εσείς. Γιατί σαφώς θα είναι πολύ ευαίσθητες οι συζητήσεις σε επόμενες μέρες και εβδομάδες. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τις απόψεις σας. Δεύτερον, για την χρηματοδότηση. Η δικαιωτική χρηματοδότηση οπωσδήποτε πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όπως σωστά επισημάνατε υπάρχουν πάρα πολλά έργα, ειδικά στον τομέα της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας, αλλά πρέπει να αποδίδουν για να επενδύσουν οι ιδιώτες επενδυτές. Πώς δηλαδή θα γίνει το σχέδιο Juncker ε, τελείως ε, μη γραφειοκρατικό για να εκμεταλλευτούμε ακριβώς τα κεφάλαια που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν κεφάλαια και έργα, το θέμα είναι πού θα συναντηθούν. Το αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες λεπτομέρειες συγκεκριμένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Βεβαίως το πρόβλημα πάντα είναι ποιος ε, θα μιλήσει πρώτος. Στην Ήτρε η πράσινη είναι περισσότερη, οπότε ο κύριος ε, Τούρμες, Κλοντ Τούρμες έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτή την γενικότερη παρουσίαση του τι μας ε, περιμένει. Προσωπικά θα προτιμούσα η Κομισιόν να το πει αυτό ενεργειακή και κλιματική ένωση γιατί αφορά βεβαίως και την περιβαλλοντική διάσταση. Εγώ σοκαρίστηκα πριν από 1,5 μήνα όταν είδα μια διαρροή ε, και δεν έπαιζαν κανένα ρόλο οι πολίτες. Και τώρα μας λέτε πως το αντιμετωπίσατε αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε μια ενεργειακή κλιματική ένωση χωρίς τους πολίτες και τις ε, πόλεις. Χρειάζεται μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και έχετε μια σχετική πρόταση και αυτό είναι θετικό. Για την Ρωσία οφείλω να πω πως ε, προσωπικά σοκαρίστηκα από την υποδοχή που είχατε στην Μόσχα. Νομίζω πως όσοι σας ξέρουν λίγο γνωρίζουν πως είστε άνθρωπος ήρεμος, συμφιλιωτικός και ήταν σκληρό αυτό που σας έκαναν. Η ανάλυση μου εδώ και 1,5 χρόνο λέει πως υπάρχει μόνο μία απάντηση στην Ρωσία. Η Ευρώπη να πάει για έναν στόχο αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας 40%. Έτσι θα εξοικονομήσουμε ένα 40% της ενέργειας και έτσι θα δημιουργήσουμε ασφάλεια και θα ξέρουν όσοι μας πουλάνε ε, αέριο, πώς θα πρέπει να γίνει και με άλλους οικονομικούς όρους. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την πλευρά της ε, ζήτησης και βεβαίως ε, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το σημαντικότερο και λιγότερο γραφειοκρατικό μέσο, ο οικολογικός σχεδιασμός για να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές και να μειωθεί η ζήτηση ηλεκτρισμού. Πρέπει λοιπόν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Για τις ανανεώσιμες κάποιοι συνάδελφοι λένε πως είναι ακριβές. Ε, συγγνώμη, κάνετε λάθος. Ήταν ακριβές. Το κόστος που έχουμε δει στα φωτοβολταϊκά είναι εντυπωσιακό. Ήμουν πρόσφατα σε μια διεθνή διάσκεψη όπου έχουμε φωτοβολταϊκά για, με 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην Αφρική που υπάρχει ήλιος. Οπότε είναι φτηνότερο από άλλες επιλογές. Το θέμα είναι για εμάς πως έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Η Ρωσία έχει δώσει 25 δισεκατομμύρια πιστώσεις με μηδενικό επιτόκιο στην βιομηχανία των φωτοβολταϊκών που ανταγωνίζεται με τη δικιά μας. Ο Αμερικανικός στρατός αφού έχασε δεκάδες στρατιώτες κατά τη μεταφορά δίζελ στο Αφγανιστάν ε, αναζητά νέες πηγές ε, μέσω της φωτοβολταϊκής, το ίδιο και η πολιτεία της Νέας Υόρκης που δίνει 750 εκατομμύρια ευρώ. Εάν θέμε λοιπόν ε, οι ανανεώσιμες να γίνουν νούμερο ένα, χρειάζεται μια, μια διάσταση βιομηχανικής πολιτικής που θα δώσει μια απάντηση σε αυτές τις επιθέσει επιθέσεις περί χρηματοδότησης. Τέλος, η περιφερειακή διακυβέρνηση είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. 73% των πολιτών μας θέλει μια ενεργειακή ε, ένωση, ενώ ε, τα κράτη λένε μην ασχολείστε με το ενεργειακό μας μείγμα. Οπότε αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε μόνο στο περιφερειακό επίπεδο. Αν μπορείτε λοιπόν να μου δώσετε κάποιες ε, λεπτομέρειες για την νοτιοανατολική Ευρώπη, γιατί εκεί πέρα νομίζω χρειάζεται αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο κύριος Νεοκλής Ηλικιώτης. Ε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε αναλάβει όντως ένα δύσκολο έργο, αυτό της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Κατά την άποψή μας, για να μπορέσει η τέτοια ένωση να λειτουργήσει θετικά, είναι σημαντικό να τεθεί στο επίκεντρο ο πολίτης, ο καταναλωτής, οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μας η ενέργεια είναι βασικό ανθρώπινο αγαθό σήμερα και είναι σημαντικό μέσω τη Ενεργειακή Ένωση να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Γιατί κύριε Αντιπρόεδρε υπάρχουν αρκετοί πολίτε σε πολλές περιοχές της Ευρώπης σήμερα ε, που είναι πραγματικά ε, στην ενεργειακή φτώχεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να συμβάλλει η Ένωση ώστε να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση για όλους φθηνής ενέργεια. Είναι σημαντικό επίσης ε, για μας να διασφαλιστεί πω τα κράτη θα έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο θα υπάρχει δηλαδή δημόσιος έλεγχος αλλά και δημόσιες ε, υποδομές. Η Ενεργειακή Ένωση, ε, επειδή αναφέρθηκαν κι άλλοι συναδελφοί, πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι το συγκεκριμένο σήμερα. Ένα ακόμα ε, θέμα είναι η άρση της απομόνωσης των κρατών. Κύριε Αντιπρόεδρε, γνωρίζετε ότι έχει τεθεί ο στόχος να υπάρξει μέχρι τέλος του 2015 και δεν βλέπουμε να μπορεί να είναι υλοποιήσιμος αυτός ο στόχος για να έρθει απομόνωση κρατών και περιεχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Και για μας επίσης είναι σημαντικό να, να ακούσουμε προτάσεις πιο συγκεκριμένες για την πρόθεση της συνεργασίας με τα γειτονικά μας κράτη με στόχο και την ειρήνη αλλά και την οικονομική ευημερία των λαών και γι' αυτά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα ε, το τι μέτρα πρέπει, ε, μπορούν να ληφθούν στα πλαίσια τη Ενεργειακή Ένωση. Τέλο, επειδή γίνεται αναφορά σε εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, θα ήθελα να υπογραμμίσω ξανά ότι στο πλαίσιο τη Ευρω... Ευρω... Ε, Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στρέψει την προσοχή της και στα κοιτάσματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και σε έναν κράτος αλλά και στις χώρες της περιοχής είναι μια πορεία εναλλακτική ε, η να εγκαθιδρυθεί ένας διάδρομος από την Ανατολική Μεσόγειο για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την παρουσία της ε, και πολιτικά αλλά και με τη χρηματοδότηση συνέργων σε αυτήν την περιοχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σαφχάουζερ από τους μία γραμμένους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και με συγχωρείτε γιατί θα πρέπει να φύγω γιατί έχουμε ταυτόχρονα και συνεδρίσει της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να πω το εξής. Κύριε Επίτροπε, όπως η Ευρώπη προσπάθησε να υποστηρίξει την ε, οικονομική ανάπτυξη, αλλά τελικά προκάλεσε την ύφεση. Με την ενεργειακή ασφάλεια, όπω προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να, μήπως τελικά προκαλέσουμε την ενεργειακή ανασφάλεια. Εγώ ξεκίνησα ως διευθυντής ε, του ενεργειακού στην Αλσατία, με μακροχρόνιες συμβάσεις με εξασφαλισμένες τιμές που επέτρεπαν την ε, μακροχρόνια προβλεψιμότητα. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε διαφάνεια για να προτιμάσουμε τις κατάλληλε επενδύσει. Η αγορά των σπότ, η αγορά, την, η ανοιχτή αγορά ε, δημιούργησε προβλεψιμότητα αλλά ε, όχι έτσι όπως την προτείνατε εσείς με την ενεργειακή ασφάλεια που ε, υπονοείτε. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την επικουρικότητα. Είναι ε, μάταιο να θέλουμε να δημιουργήσουμε ενεργειακή ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν υπάρχει ήδη σε εθνικό επίπεδο, σε επικουρικο... στο επίπεδο τη επικουρικότητα. Και η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει με την ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι ένα αγώνα πολύ σημαντικό για μένα. Μιλήσατε για 20%. 20% θα πει 80 δι. 80 δι θα πει 800 δι επενδύσει. Ο πρόεδρο μπουζ ζήτησε να ε, παραμείνουμε στη λογική του προγράμματος Juncker για να συμμετέχουμε και να αντλήσουμε όλες αυτές τις επενδυτικές προσπάθειες για την ενέργεια. Αλλά η ποσοτική χαλάρωση για τις ε, τράπεζες. Τα χίλια δις δεν θα έπρεπε να γίνονται για τις τράπεζες αλλά για την πραγματική οικονομία. Ώστε την πραγματική οικονομία να αναθερματεί. Αυτό θα τα άλλαζε όλα άρδιν. Δεν, μην αυταπατώμεθα διότι λέτε ότι υπάρχουν αρκετές επενδύσεις. Εδώ και 20 χρόνια ακούω ότι έχουμε αρκετές επενδύσεις αλλά στην πράξη τίποτε δεν γίνεται. Οι εταιρείε ενέργεια δεν έχουν αρκετά κεφάλαια για να μπορέσουν ακριβώ με την ενεργειακή αποδοτικότητα να έχουν και την απαραίτητη απόδοση. Αυτά τα τρία ερωτήματα θα ήθελα να απαντηθούν. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Oh, Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο κύριος Χέλμερ. Από την Ευρώπη της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Συχνά παραθέτω τα λόγια του συναδέλφου Ταγιάννη, που όταν ήταν Επίτροπος Βιομηχανίας έλεγε ότι οι ενεργικές τιμές δημιουργούν βιομηχανική βιομηχανικό μακελιό στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι και εσείς το αναγνωρίζετε αυτό. Και εδώ προετοιμαζόμενος για αυτή τη μεγάλη ομιλία ε, σκέφτηκα να διερευνήσω τις εκτάσεις αυτού του βιομηχανικού μακελιού και συνείδησα μέλη από τα δηληστήρια πετρελαίου, από τη χαλιβουργία και από την βιομηχανία του σιδήρου στην ε, Ευρώπη. Έχουν χάσει το 40% των δυνατοτήτων του τα τελευταία 7 χρόνια. 40.000 ε, θέσει εργασία έχουν χαθεί. Η ζήτηση αυξάνεται όμω, δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί και δυστυχώ καλύπτεται από εισαγωγέ, πάνω από το 50%. Ε, παρόμοια τα στοιχεία για τον Χαλβά, όπου έχουν χαθεί 50.000 εργασία, έχουν κλείσει εργοστάσια. Το ίδιο και για τα δηληστήρια πετρελαίου. Είναι φτηνότερο να φέρει κανεί ε, πετρέλαιο που έχει δηληστεί στην Αφρική, τη Ρωσία από ότι να περάσει εδώ στη δίληση. Άρα ε, κλείνουν τη ληστήρια και 10.000 ε, θέσεις εργασίας άμεσες, 4.000 έμεσες. Αυτό είναι το μακελιό που έχουμε προκαλέσει. Ε, ας μην πιάσω τώρα και την ιαλουργία, το, το τσίμεντο βιομηχανία και τη χημική βιομηχανία. Παρόμοιες ιστορίες θα βρούμε και εκεί να ψάξουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε βιομηχανίες ε, που καταναλώνουν πολλή ενέργεια, που έχουν γαντζωθεί με τα νύχια για να σωθούν και την ίδια στιγμή το Κοινοβούλιο μιλά για το απόθεμα της ενεργειακής σταθερότητα. Εδώ ο στόχος είναι να αυξηθούν και άλλο οι τιμές και η Ευρώπη να γίνει ακόμα λιγότερο ανταγωνιστική για να μπορεί κανείς να ασκήσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν κρίσιμη σημασία σημείο κύριε Επιτροπέ. Από την πετρελαιοβιομηχανία έχω αντίτυπο μιας έκθεσης της Βρετανικής κυβέρνησης η οποία αναφέρει ότι οι εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα που σχετίζονται με το εισαγωγής πετρέλαιο που έχει δηληστεί είναι 45% περισσότερες από ότι το πετρέλαιο που, από το πετρέλαιο που προηγουμένω το δηλίζαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αποδεκτικά στοιχεία από την Χαλιβουργία λένε ότι ο εισαγμένο χάλιβα σημαίνει διπλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από την ποσότητα που είχαμε προηγουμένω στην Ευρώπη. Άρα η πολιτική μα είναι να εξάγουμε θέσει εργασία, να εξάγουμε τι επενδύσει, να εξάγουμε την επεξεργασία των προϊόντων και να αυξάνουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ταυτόχρονα. Κύριε Επίτροπε, εάν αυτό δεν είναι καθαρή τρέλα, τι είναι. Σα uh, Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Αντιπρόεδρε, εάν θέλετε, δώστε μας τις απαντήσεις και παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να τα διατρέξω όπως ε, ε, τα θέσατε, κύριε Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Είναι επίκαιρη και θα συνδυαστεί και με τις δικές μας εργασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τη μελετήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε από την έκθεση. Ε, όσο για τη Ρωσία, ε, ένα θέμα που είναι ήδη επιτάπητος, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι περίπλοκος και πολύ δύσκολο στη συμπεριφορά αυτός ο εταίρος. Το έχω πει επανειλημμένος. Για μια τέτοια εταιρεία όπως η Gazprom, ο καθιερωμένος τρόπος επικοινωνίας είναι να μιλά κανείς στους ε, πελάτες και τις χώρες των οποίων οι εταιρείε έχουν συμβάσεις με την Gazprom. Εκεί θα χρειαστούν ριζικέ ε, αλλαγέ και ανακοινώνονται ένα δεκαπενθήμερο. Αυτό δεν είναι η καθιερωμένη συμπεριφορά. Έχει να κάνει με το ότι αν η Γκάσπρομ είναι ή όχι αξιόπιστος προμηθευτή αερίου. Εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα αναγκαστικά. Ε, μετά την επίσκεψή μου στη Μόσχα, ε, νομίζω όχι μόνον εγώ εξεπλάγει, αλλά και άλλοι συνάδελφοι με, τον Ρώσο εταίρο που, με τους Ρώσους εταίρους που συναντήσαμε. Διότι φαίνεται να ήταν ριζική η μετατόπιση της αντίληψής τους ε, στο πώς θα προμηθευόμαστε αέριο στο μέλλον. Ένα σύστημα που προτείνουν και απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Υπάρχουν ε, μακροπρόθεσμες συμβάσεις εδώ, μακροχρόνιες συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, αλλά δεν αφορούν μόνο τον όγκο αερίου, αλλά και το σημείο της προμήθειας. Και σίγουρα δεν είναι τα τουρκοελληνικά σύνορα αυτά, ε, αυτά τα σημεία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για προμήθεια, για λυσίδες, για συμβάσεις που έχουν σαφείς ρήτρες για τα θέματα αυτά. Όμως παραμένει αναλύτω το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε διαρκώς αυτό το πρόβλημα άγχους. Διότι το θέμα είναι, δεν είναι μόνο τι θα γίνει το χειμώνα και πώ θα γίνουν σεβαστέ οι συμφωνίε του χειμώνα, αλλά τι θα γίνει και το καλοκαίρι. Εκεί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Οι Ρώσοι εταίροι φαίνεται να υποστηρίζουν ότι μετά το τέλο Μαρτίου θα επιστρέψουν στι συμβάσει που ίσχυαν πριν την κρίση στην Ουκρανία. Αυτό θα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, διότι αυτό ήταν το ερώτημα του κύριου Κάριντς. Νομίζω ότι σαφώς πρέπει να δουλέψουμε όλες τις διαστάσεις. Βεβαίω πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προμήθεια, όχι μόνο τι οδού προμήθεια, αλλά και τι πηγέ του αερίου. Τον Φεβρουάριο είναι ένα σημείο ρώσιμο για μας από αυτή την προοπτική, διότι θα συζητηθεί το τι θα γίνει με τον, ε, με τον νοτιοανατολικό διάδρομο. Έχουμε πολύ σημαντική συνάντηση λοιπόν ε, με τις εκπληρώσεις των χωρών από τις οποίες θα περάσει ο νότιος διάδρομος αλλά και με τους Ρώσους διότι μετά τον Αμπούκο και τι πολιτικέ προτεραιότητε που έχουμε, με την πολιτική προβολή που θέλουμε να του δώσουμε, του μηχανισμού με του οποίου θα δημιουργήσουμε πάλι ένα οδικό χάρτη, θα δούμε πώ πρέπει να προχωρήσουμε για να δημιουργήσουμε το νέο αγωγό. Τι προβλήματα πρέπει να επιλύσουμε ώστε να καταλήξουμε σε, επιτυχή, σε επιτυχές πέρας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με το hub, το κομβικό σημείο αερίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε στη Μεσόγειο. Ε, για το θέμα αυτά. Πολλά μπορούν να γίνουν ε, με την Αλγερία και θα πρέπει να ξαναδούμε και το υγροποιημένο αέριο. Έχουμε ήδη σαφείς δυνατότητες στην Ευρώπη, αλλά και πάλι δεν τις αξιοποιούμε πλήρως. Δεν έχουμε σαφείς διασυνδέσεις, ώστε το υγροποιημένο φυσικό αέριο να αξιοποιείται πιο εντατικά. Άρα, μια από τις ιδέες που θα προτείνουμε είναι να υπάρχει μια συνολική ε, θεώρηση για την ε, ενεργειακή μας στρατηγική. Να δούμε πώς μπορούμε να μοιραστούμε τους πόρους, τις δυνατότητες υγροποιημένου αερίου. Όχι μόνο με παζάρεμα, αλλά με μια πολιτική ασφάλισης ώστε να σταθεροποιηθούν όσο γίνεται αυτέ οι περίπλοκε τιμέ του αερίου. Και επίση συμφωνώ ιδιαίτερω μαζί σα ότι όταν μιλάμε για τι διακυβερνητικέ πια συμφωνίε πρέπει να το δούμε το θέμα διαφορετικά. Ορθώ είπατε ότι έχουν υπογραφεί και μετά ε, παρουσιάζονται στην Επιτροπή για να αναλυθούν, να δουν αν, να δει η Επιτροπή αν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφανέστερη η διαδικασία εάν τα κρατημέλη ήταν ανοιχτότερα και διαφανέστερα για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων των ε, συμφωνιών αυτών. Θα έπρεπε να είναι μέλο τη διαπραγματευτική ομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία τέτοιων διαστάσεων υπογράφεται να έχουμε βεβαιωθεί από πριν ότι συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Να μην υπάρχουν εκπλήξει τον για τον άλλο. Δηλαδή αυτό θα αυξήσει και τη διαπραγματευτική δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει τι διαπραγματευτικέ θέσει των κρατών μελών και των εταιριών μα όταν ε, θα διαπραγματεύονται. τις ε, ενδεχόμενες συμφωνίες. Κοινέ αγορές αερίου. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Ένα θέμα πολύ τεχνικό. Ένα θέμα που απαιτεί ενδελεχή νομική εξέταση. Ε, έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις εδώ. Οι δυτικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αγορά που λειτουργεί εύρυθμα, με τους μηχανισμού τη αγορά να εφαρμόζονται χώρες που πιστεύουν ότι πρέπει να θεθούν ελεύθερες οι εταιρείε να λειτουργούν και να μην πειράξουμε το σύστημα. Είναι μία ομάδα, αλλά στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Εκεί, βασισμένοι στις εμπειρίες του παρελθόντος, θα προτιμούσαν να έχουν τη δυνατότητα να υπάρχουν κοινέ αγορές αερίου, διότι μεμονωμένα αγοράζουν μόνο μικρέ ποσότητε αερίου. Θα είχαν καλύτερε τιμέ λοιπόν αν αγοράζαν περισσότερο και αν από κοινού. Άρα αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μήπω πρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά το θέμα αυτό και το μελετούμε εντελεχώ. Υπάρχουν δύο πολιτικέ προσεγγίσει βλέπουμε και πολλέ προκλήσει από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού, από την άποψη τη ε, συμβατότητα της προσέγγισης με τους κανόνες του ΠΟΕ ε, και τις υποχρεώσεις που, ε, που πηγάζουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ. Και επίσης τη δυνατότητα της ε, εθελοντικής συνάθρησης των αγορών το πόσο μπορούμε να πυροδοτήσουμε ένα μηχανισμό όταν η κατάσταση είναι δυσχερή, μη διαφανής ή όταν βρισκόμαστε σε κρίση. Αυτή είναι η συλλογιστική μα. Αναλύουμε όλε αυτές τις πτυχέ όπως σα τι ανέφερα και είναι ένα θέμα που θα απαιτήσει περαιτέρω προσπάθεια και μελέτη. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στις ερωτήσει του κυρίου Νίκα για τους ευάλωτους καταναλωτές. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα εδώ είναι ότι αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι υπάρχει πρόβλημα. Διότι θα ξέρετε ότι έχουμε διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ε, εάν ρωτήσετε διαφορετικούς φορείς ή ε, εταιρείες των ε, κρατών μελών, των κρατών μελών, θα σας δώσουν διαφορετικούς αριθμούς με διαφορετικά ποσοστά. Αυτό περιπλέκει την συνολική θεώρηση και την αναζήτηση λύσεων. Όμως, εάν αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι ήδη σημαντικό. Υπάρχουν Ευρωπαίοι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη θέρμανση, δεν μπορούν να πληρώσουν την, το λογαριασμό του ηλεκτρικού, της ενέργειας. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όμως νομίζω ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα ενεργειακής πολιτικής, αλλά και κοινωνικών πολιτικών. Είναι ε, ένα θέμα που να το δούμε από κοινό με την Επίτροπο Τάισεν. Και το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο κρατών μελών. Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε όλα αυτά να λυθούν. Ε, αναφερθήκατε, νομίζω, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Πρέπει να στηρίξουμε το όλο πρόγραμμα. Θα μειωθούν οι λογαριασμοί για τα νοικοκυριά. Θα ε, μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου ε, του άνθρακα και θα βελτιωθεί η κατάσταση και, για τα, και σε περιφερειακό επίπεδο. Πολλοί δήμαρχοι μας είπαν ότι χρησιμοποιούμε ένα νέο σύστημα με αγορές κοινέ για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ε, τους δημόσιους χώρους, οπότε και εμείς εξοικονομήσαμε χρήμα, αλλά αυτό εξυπηρετεί και τις εταιρείες ως δημοτικές αρχές. Ε, αν όμως πρέπει να γίνει αυτό σε επίπεδο ιδιωτικών οικοκυριών, σε επίπεδο μεγάλων συγκροτημάτων ε, κατοικιών. Εδώ χρειάζονται περισσότερα χρήματα, περισσότερη λεπτομέρεια. Θα είναι πολλά ε, αυτά που θα πρέπει να γίνουν και εξαρτάται από το να βρίσκεται κανεί σε μια μικρή ή μεγάλη κοινότητα, ένα μικρό ή μεγάλο δήμο. Ε, πρέπει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο, τον κύριο Χόγερ, για να δούμε ε, τα παραδείγματα και από τη Ρουμανία και το κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο εργαλείο εύχριστο για τις δημοτικές αρχές σε όλη την Ευρώπη που να λέει αν θέλετε μια τέτοια, ένα τέτοιο πρόγραμμα, ιδού οι συμβουλές, ιδού η δυνατή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Juncker ή από τους θεσμικούς επενδυτές που μπορεί να ενδιαφέρονται και να μπορούμε να βοηθήσουμε για την απαλυθή αυτών των αρχικών δυσκολιών των τόσων λεπτομεριών και των αποτρεπτικών στοιχείων ότι είναι πολύ δύσκολο για να γίνει. Αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στην προσέγγιση των ευφυών πόλεων. Ε, διότι έχουμε την ενεργειακή αποδεκτικότητα για τα σπίτια, ε, για τι μεταφορέ. Έχουμε πρόβλημα με τι υποδομέ και έχουμε 80% των Ευρωπαίων σε αστικά κέντρα. Πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα με τι πόλει. Αλλά το ζήτημα είναι υπαρκτό και νομίζω θα το ξαναδούμε σύντομα ε, για να βρούμε τη σωστή ισορροπία και από την πλευρά τη επικουρικότητα από τη μια ε, υποστηρίζω τους ε, δημάρχους, τους 600 δημάρχους που εργάζονται βάσει του Συμφώνου των ε, Δημάρχων, από την άλλη, χρειάζεται και ευρωπαϊκό συντονισμό και συνεργασία και νομίζω και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα ακούσουν του δημάρχου και θα στηρίξουν τι προτάσει του. Ένα άλλο ζήτημα. Ναι, ο πρόεδρος Μπούζεκ μου λέει πρέπει να είμαι συντομότερος, θα προσπαθήσω. νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ένδυα, την ε, ευάλωτη κατάσταση και τις ε, τιμές του ηλεκτρικού που αναφέρατε, το ανέφεραν πολλοί οι βουλευτέ, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το σχεδιασμό της παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είδατε στις διαφάνειες πόσο στηρίζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ξαναδημιουργούμε ε, στην ενεργειακή αγορά εθνικά σύνορα δημιουργήσαμε τεχνητούς φραγμούς, ε, τεχνικές δυσκολίες. Αυτό μας ξαναπήγε στο σημείο 0. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε την αγορά του ηλεκτρικού στην ε, Ευρώπη. Πώς μπορούμε να έχουμε εξοικονομήσει κλίμακας, τι μηχανισμούς μπορούμε να έχουμε για την αγορά, τι σχέδια στήριξης. Ξεκινήσαμε νομίζω σωστά με την έγκριση των νέων κανόνων για την κρατική βοήθεια για τις ανανεώσιμες πηγές. Εκεί βλέπουμε πώς θα μπορούσε να προχωρά αυτή η διαδικασία και πώς σταδιακά θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παράγοντες που λειτουργούν στην αγορά να συμπεριληφθούν στην αγορά διότι όπως είπατε μειώνεται η τιμή των ανανεώσιμων και μειώνεται δραματικά. Σύντομα θα είναι ανταγωνιστικές και θα είναι ε, ένα από τα στοιχεία τα κανονικά της αγοράς. Θα επηρεάσει αυτό την ενέργεια συνολικά. Πολλοί από εσά είπατε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Συμφωνώ απολύτως. Χωρίς ευφυή δίκτυα χωρίς ε, διασυνδέτες που θα μας επιτρέπουν την ε, ελεύθερη ροή ενέργειας στην Ευρώπη δεν μπορεί να χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Πρόσφατα ένας ε, διευθυντής εταιρεία μηχανικής μου είπε ότι αν σήμερα παρκάρει κανείς πέντε ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ένα δρόμο, μπορεί να, σε μια οποιαδήποτε οδό, μπορεί να προκαλέσει blackout σε όλη τη γειτονιά. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τι υποδομέ μα, να γίνουν ευφιέστερα τα δίκτυά μα. Αυτό να μην συμβαίνει. Εάν θέλουμε να δώσουμε δύναμη στους καταναλωτές, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνουν την πληροφορία που χρειάζονται για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Ότι μπορούν να κάνουν την μετατόπιση ενέργειας. Εκεί χρειάζονται επενδύσεις λοιπόν στις υποδομές, όντως. Και γι' αυτό Συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο ότι πρέπει να παρακολουθούμε τα σχέδια περί υποδομών και να τα ε, στηρίζουμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα με τους αγωγούς. Ένα από τα διευθυντικά ταμεία για τα νέα κράτη-μέλη. Ένα σχέδια κοινού κοινής ωφελίας που συνδέονται με την ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική. Μετά έχουμε το πρόγραμμα του Εργαλείου για τη Διασύνδεση της Ευρώπης και μετά έχουμε και το πρόγραμμα Juncker για τις επενδύσεις. 72 προγράμματα ενέργειας εξετάζονται την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και είναι όριμα για εφαρμογή. Όμως, εάν ρωτήσει κανείς την απλή ερώτηση, τι μπορεί να κάνει κανείς για αυτή τη χώρα τώρα, όπως έγινε με την Βουλγαρία και την κατάργηση, την ανακοίνωση της κατάργησης του South Stream. Ε, εδώ όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα, μαζί. Άρα πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσουμε να βελτιώσουμε τις σωστές ε, πληροφορίες, να τις συνδυάζουμε με τρόπο διαφανή, να ξέρουμε ποια ε, προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτηθούν πρώτα. Να υπάρχει μια αποτίμηση, αλλά αυστηρή. Διότι πολλέ χώρε παραπονούνται ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Εάν είχαν του διασυνδέτε, όπω του είχαμε προτείνει, θα ήταν σε πολύ διαφορετική κατάσταση σήμερα. Δεν είναι λοιπόν θέμα δημιουργία ευκαιριών, αλλά και πώ θα ε, ελέγχουμε, πώ θα παρακολουθούμε και θα βεβαιωνόμαστε ότι γίνονται όσα πρέπει δεν είναι μόνο θέμα ενεργειακής ασφάλειας για ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά είμαστε τόσο αλληλέμπετοι μεταξύ μας στις ανάγκες μας, που ένας να λείπει από τους διασυνδέτες, καταραίει όλο το σύστημα. Ολόκληρη περιοχή. Για τις διασυνδέσεις αυτές καθ' αυτές. Όπως εξήγησα, τι θέλουμε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, και εδώ θα ολοκληρώσω γιατί ο πρόεδρος με κοιτάει στραβά, με κοιτάει αυστηρά, όχι, όχι, απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ήταν ε, πολύ σημαντική ερώτηση του κυρίου Σιλικιώτη και άλλων. Ε, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αυτό που θέλουμε να σας ε, παρουσιάσουμε είναι το εξής. Ενεργειακή Ένωση, στρατηγική για το κλίμα και οδικός χάρτης για το πώς θα οδεύσουμε πώ θα φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή, την Ενεργειακή Ένωση, στα πέντε τουλάχιστον πρώτα χρόνια βάσει τη εντολή μα. Και θέλουμε και έναν οδικό χάρτη για το Παρίσι. Ποια θα είναι η διαπραγματική μα θέση για το Παρίσι. Διότι ξέρω ότι όλα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ και είναι αλληλένδετα. Οι τρει διαστάσει ε, που ανέφερα προηγουμένω ε, είναι αλληλένδετε με τη διαπραγματική μα θέση όπω θα την εκφράσουμε στο Παρίσι. Και επίση θα θέλαμε και μια ανακοίνωση για το πώ θα πετύχουμε τι υποχρεώσει μα αυτές που συμφωνήσαμε για το 10% διασύνδεσης μεταξύ όλων των κρατών μελών μέχρι το 2020. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικότατο έγγραφο που θα προσανατολίσει τη συλλογιστική και την εργασία μας στο μέλλον. Για τα προγράμματα υποδομών. Ο κύριος Πέτερσεν ρώτησε και είναι αντιπρόεδρος, οπότε οπωσδήποτε πρέπει να απαντήσω στην ερώτησή του. Τι μπορούμε να κάνουμε με την νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί, που είναι πολύ σωστή, αλλά δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να είμαστε αυστηρότεροι, νομίζω. Πολύ αυστηρότεροι στο πώ παρακολουθούμε την εφαρμογή. Πώ ελέγχουμε, πώ επιμένουμε για την μεταφορά. Αυτό που προτείνουμε τώρα είναι διάλογο, λεπτομερέστερος διάλογο υλοποίηση με τα κράτη-μέλη. Όταν κοιτάζουμε τι νομοθεσία ισχύει, και εάν ή γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά, πρέπει να δούμε αν το ζήτημα είναι πολιτικό, οικονομικό, εάν υπάρχει πρόβλημα με του εμπειρογνώμονε ή την τεχνογνωσία σε επίπεδο κράτου μέλου, πώ αντιμετωπίζεται. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Πώ θα προχωρήσουμε με τα προγράμματα υποδομή, πώ επενδύουμε στου διασυνδέτε. Να ρωτήσουμε εάν χρειάζονται τη βοήθειά μα τα κατημέλη, εάν μπορούμε να προοδεύσουμε με τη συνδρομή όλων. Διότι η αλήθεια είναι το τρίτο ενεργειακό πακέτο είναι πολύ σημαντικό, αλλά η μεταφορά και η υλοποίησή του ως τώρα είναι σαφώς ε, πλημελής. Δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική και πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπαθίες μας. Τελευταίο που θέλω να πω για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πολλοί από εσά ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. και την ανακοίνωση για το Southrim. Νομίζω ότι είναι πολύ απλή απάντηση. Χρειάζεται νέο ε, βασικό σχέδιο για την Ανατολική Ευρώπη και τη διασύνδεσή της με την κεντρική. Άρα, αποφασίζουμε ότι θα υπάρξει υψηλό επίπεδο ομάδα που θα συζητηθεί, ε, που θα συναντηθεί πρώτη φορά στις 9 Φεβρουαρίου. Η Πρωθυπουργό τη Βουλγαρία θα δείξει την αλληλεγγύη της στην πρώτη, με την παρουσία τη στην πρώτη συνάντηση και θα δει σε πρώτη φάση ομάδα αυτή τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε με τη διαφοροποίηση τη προμήθεια αερίου και πώ μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε στη συνέχεια για την ηλεκτρική ενέργεια ότι υπάρχουν ε, οι απαραίτητοι διασυνδέτε. Πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή πώς σε αυτό το μέρος της Ευρώπης μπορούμε να έχουμε καλύτερη ένταξη στα ενεργειακά δίκτυα της Ενεργειακής Ένωσης και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως μετά τις εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος. Κύριε Πρόεδρε, εδώ ολοκληρώνω. Δώσετε όλες τις απαντήσεις, διότι όλοι οι βουλευτές πρέπει να ικανοποιηθούν. Μία ή δύο προτάσεις, αν θέλετε, τις έχετε. Με συγχωρείτε, κύριε Αντιπρόεδρε σύντομα, αλλά ικανοποιήστε όλους. οικολογικό σχεδιασμό και βιομηχανική πολιτική, νομίζω ήταν ε, η ερώτηση του κ. Χέλμερ. Για τον οικολογικό σχεδιασμό, Ίσως τέθηκε από δύο διαφορετικές ε, φωνές αλλά από διαφορετικές παρατάξεις. Ε, για τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει να μας βοηθήσετε να επικοινωνούμε για τον οικολογικό σχεδιασμό όπως πρέπει. Ε, η ουσία είναι πώς θα διαμορφώνεται και η κοινή γνώμη. Είναι απολύτω απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και καταστρέφει τι προσπάθειέ μα για ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρέπει απλούστατα να πούμε στου πολίτε ότι χάρη στον οικολογικό σχεδιασμό και τη σχετική οδηγία, μέχρι το 2020 θα έχουμε ε, ε, την ίδια ε, κατανάλωση ενέργεια όπω στην Ιταλία μέσα σε ένα χρόνο. Βλέποντα του στόχου τη ενεργειακή αποδοτικότητα του 20% μέχρι το 2020, σήμερα μόνο το μισό, το 9%, το, 9% το πετυχαίνουμε χάρη στην οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Οι καταναλωτέ το θέλουν αυτό. Είναι κάτι που του ε, χαμηλώνει και του λογαριασμού ηλεκτρικού και είναι καλό και για τη βιομηχανία γιατί δεν πρέπει να περνάνε τη δικασία πιστοποίηση για κάθε κράτο μέλο ξεχωριστά. Άρα έχουμε μια νέα αγορά εδώ και αυτό λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που προσπαθούμε είναι να βελτιώσουμε την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ώστε να γίνει διαφανέστερη, λιγότερο παραγματική και να βασίζεται στα πρόσφατα στοιχεία. Όμω νομίζω ότι πραγματικά το εργαλείο αυτό το χρειαζόμαστε για να είμαστε βέβαιοι ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, ισχύει και για τις ηλεκτρικές ε, συσκευές. Και ε, σε ό,τι φορά την βιομηχανία, πολλοί είναι εκείνοι που μίλησαν για τους βιομηχανικούς κλάδους που καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Μεγάλη πρόκληση αυτή για όλους μας, αλλά νομίζω ανέκαθεν προσπαθούσαμε να βρούμε μια σωστή λύση. Ε, μιλήσαμε και προτείναμε τις διατάξεις διαρροής άνθρακα ε, για να προστατευτούν οι ενεργειακά εντατικές βιομηχανίες από τις ενδεχόμενε διαρροές. Αλλά νομίζω αν μιλάμε για ε, τιμές του ηλεκτρικού, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αγορά, να δημιουργηθεί εσωτερική αγορά με των φραγμών, με αλλαγή του σχεδιασμού του ηλεκτρικού τοπίου και με το εργαλείο σταθεροποίησης της αγοράς ε, με αναθεώρηση του συστήματος ανταλλαγής δικαιωμάτων ε, ε, εκπομπών ώστε να έχει μια εικόνα ο επιχειρηματικό κόσμο και η κοινωνία και για την περίοδο μετά το 2020. Εάν άκουσα πάντω κάτι από τον οποιονδήποτε εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κόσμου μετά από τι συνομιλίε που είχα όλο αυτό το διάστημα, ένα πράγμα θέλουν πριν επενδύσουν. Ρυθμιστική σταθερότητα μου είπαν, εάν αυτό μας το εξασφαλίσετε, εάν μας εγγυηθείτε ότι θα υπάρχει ρυθμιστική ε, σταθερότητα, ε, νομοθετική σταθερότητα με τις προτάσεις σας, ευχαρίστως να πάμε στην κατεύθυνσή σας. Για μας είναι συμφέρον ε, να είναι τα προϊόντα μας ενεργειακώς αποδοτικά, φιλικά προς το περιβάλλον, να εξοικονομούν ενέργεια για τους πελάτες μας. Βεβαίως, θα τα πουλάμε και στο εξωτερικό. Θα είναι το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας επιτρέπει να διαφημιστούμε στο εξωτερικό. Είναι νέε ευκαιρίε αυτέ για τη βιομηχανία, νέε ευκαιρίε για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία στο Παρίσι, ότι θα έχουμε μια δεσμευτική συμφωνία εκεί που θα εξασφαλίσει και για την Ευρώπη και για όλους τους παγκόσμιους εταίρους ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού για τις εταιρείε μας από ό,τι ως τώρα. Καλό λοιπόν θα είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Έχουμε 17 ομιλητές. Προτείνω να κλείσει εδώ πέρα ο κατάλογος. Καταλαβαίνω πως συμφωνείτε όλοι. Ξεκινάμε Κυρία Πιλάρντε Καστίγιο Βέρα. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτς, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που αναφέρατε. Τα έξυπνα δίκτυα, τα οποία πρέπει να αναβαθμιστούν. Ξέρετε, είχαμε κάνει πολλή συζήτηση την ε, προηγούμενη φορά τελικά δεν έγινε τίποτα όπως λέτε είναι η βάση αυτό για την ανάπτυξη της ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι η διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών εταιριών δεν είναι τόσο καλή η συνεργασία και νομίζω πως πραγματικά να το βάλετε ως πραγματική προτεραιότητα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σύντομοι δεν περάσετε το 1,5 λεπτό Blanco Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει κανείς ε, με τους στόχους αυτούς. Πράγματι να μην έχουμε τόση ενεργειακή εξάρτηση, να μειώσουμε το κόστος, ε, αλλά ας περάσουμε τώρα από τις αλήθειες και τις διαπιστώσεις ε, στην ε, πράξη. Μια ερώτηση λοιπόν. Έχουμε έναν σαφές νομικό πλαίσιο που παρέχει σταθερότητα. Μιλάμε για επενδύσεις, ε, ιδιωτικές επενδύσεις βεβαίως, αλλά για ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζεται σταθερότητα. Αν δούμε την χώρα μου, Ε, βλέπετε πως ε, έτσι με τη σταθερότητα υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες. Υπάρχουν κάποιες απομονωμένες ενεργειακές νησίδες, ε, μεταξύ των οποίων και η Βυρική Χερσόνησος. Πρέπει να υπάρχει διασύνδεση και έξυπνα δίκτυα. Είναι σημαντικό αυτό για την ανταγωνιστικότητα των ε, βιομηχανιών μας. Ε, και βεβαίως κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω, το αλουμίνιο αναφέρθηκε ήδη. Έχουμε πολλά προβλήματα. Ακριβώ λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι, να μειώσουμε το κόστος. Και είναι αναγκαίο αυτό για τις ενεργοβόρες ε, βιομηχανίες. Επίσης, επίσης, θα τελειώσω. Θα ήθελα να υπάρχει κάποιο σχέδιο από την Ένωση για να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Ε, δεν είναι δυνατόν εκατομμύρια πολίτες ε, να μην μπορούν να έχουν Σας Ευχαριστώ Ουρουτσέκ για 1,5 λεπτό, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανάπτυξη του θέματος της, ενεργειακή, της Ενεργειακής Ενώσεως από τις μεγαλύτερες προσδοκίες που έχουμε είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας της προμήθειας του φυσικού αερίου. Εδώ η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Συνάδελφοί μου ήδη έθιξαν το θέμα. Εγώ θα πω ότι καθιστάμεθα μάρτυρες μια συστηματικής πολιτικής από πλευράς της Ρωσίας για να πετάξει έξω την Ουκρανία από το διαμετακομιστικό εμπόριο του φυσικού αερίου. Αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να μπει στο κέντρο των πολιτικών της Ενεργειακής Ένωσης. Έχω και μια ερώτηση για τις ανανεώσιμες τώρα. Ο τομέας των οποίων έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη λόγω των μαζικών επιδοτήσεων ορισμένες από τις χώρες που σημείωσαν πρόοδο δυστυχώς φόρτωσαν στους καταναλωτές τις τιμές, τους μετακύλησαν δηλαδή το βάρος. Εξάλλου διάφοροι λόγοι, διάφοροι λόγοι οδηγούν σε διαφορετικό δυναμικό των διαφόρων ανανόσιμων ενεργειών. Γιατί δεν συνενώνει όλες τις πολιτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χορήγηση αδειών, να ενισχύσει δηλαδή τις ε, πολιτικές αυτές στο επίπεδο της ίδιας της Ένωσης. Ευχαριστώ η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ένα βασικό θέμα. Φυσικό αέριο. και τον άξονα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Θέλω λίγο περισσότερες πληροφορίες. Η Ενεργειακή Ένωση πώς θα υλοποιήσει αυτό το gas hub, αυτό τον πόλο μεταφοράς αέριου. Μιλήσατε και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πού βλέπετε τις δυνατότητες εκεί, καθώς και τη μεταφορά του. Και τέλος, αυτή την ολιστική προσέγγιση. Κατανοώ ότι η Ενεργειακή Ένωση θα προσπαθήσει να φτιάξει μια κοινή στρατηγική από θεμάτων ενέργειας. Πώς θα γίνει αυτό για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης. Ευχαριστώ Γιούρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κάνω πρώτα μια γενική παρατήρηση. Πιστεύω ότι εάν κατορθώσουμε να φτιάξουμε μια αποτελεσματική ενεργειακή ένωση θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τώρα έχω δύο ειδικότερε παρατηρήσεις. Πρώτα, δεν υπάρχει ενιαία αγορά ενέργειας που να λειτουργεί χωρίς να μπορεί να βασίζεται σε μια ενεργειακή υποδομή. Υπάρχουν οι γνωστές ελλείψεις. Δεν υπάρχει αγωγού νεαγωγούς δηλαδή μεταξύ Ρουμανία ουτε ούτε Ουγγαρίας-Κροατίας. Αυτά είναι τα κομμάτια του μοσαϊκού που λείπουν. Αυτά πρέπει πρώτα να συμπληρώσουμε για να φτιάξουμε μια ενιαία ενεργειακή αγορά. Τώρα η διπλωματία της ενέργειας. Συμφωνώ με τον Κάρενς που είναι ο συντονιστής μας. Το να μιλούμε με μια φωνή αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να δράσει η Ένωση στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια τεράστια αγορά ενέργειας. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα τόσο πολύ από ε, προμηθευτές τρίτων χωρών. Μπορείτε λοιπόν να αναμένετε την πλήρη μας υποστήριξη στα μέτρα που έχετε ανακοινώσει. κυρία Κάλλας, ευχαριστώ. Είπατε ότι η Ενεργειακή Ένωση σημαίνει και την ελεύθερη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος και πέρα από τα σύνορα, ώστε χώρες μέλη να μπορούν να υποφεληθούν. Και το είπατε, το είπαν αυτό και άλλοι συνάδελφοι. Είπατε ότι οι διασυνδέσεις αυτές δεν θα εξυπηρετούν εμπορικούς σκοπούς, αλλά περισσότερο για να ξεπερνούνται οι εχμές, δηλαδή ε, τα σημεία όπου κινδυνεύει να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να συνδεθούν τώρα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μάλλον για να, ξε, για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός. Πώς βλέπετε να αναπτύσσεται ο ρόλος του Acer Ευχαριστώ. Α, κυρία συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε τη Επιτροπής, νομίζω η πρότασή σα είναι κρίσιμη, διότι πρόκειται για το νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης μέσα από αυτή την Ενεργειακή Ένωση. Δηλαδή, έχετε αφενός ένα τεράστιο φάσμα ως όραμα, αλλά και ταυτόχρονα ένα συγκεκριμένο δρόμο πρέπει να υλοποιήσετε. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για την τιμή του άνθρακα, δηλαδή των εκπομπών. Εάν στο δρόμο προς την συνδιάσκεψη του Παρισιού, που θέλουμε να αποβεί επιτυχής, αν στα πλαίσια του σχεδίου επενδύσεων που προωθεί ο Ζαν αν δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ορατότητα της τιμής των εκπομπών άνθρακα, όλη η παραπέρα πορεία θα αποτύχει. Χρειάζεται λοιπόν ξεκάθαρα μια παρέμβαση του νομοθέτη στην, αγορά της αγορά, στην ε, ε, της αγοράς που είναι ακατάστατη. Με τιμή για τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα που να είναι οδηγός για τις αγορές. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η τιμή του πετρελαίου. Ίσως κάτι να μην πρόσεξα, αλλά δεν νομίζω να το τονίσετε τόσο πολύ. Αφενός υπάρχει μια όθηση για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Μήπως πρέπει να προβληματιστείτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αυτό το ευεργετικό πλεονέκτημα δεν ωφελεί μόνο εκείνους που έχουν τις μεγαλύτερες δυναμικότητες, αλλά να χρησιμοποιηθεί για να προσανατολιστούν οι επενδύσεις εκεί όπου πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Βέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, πολλές ερωτήσεις σας έθεσαν και τις περισσότερες μάλιστα τις απαντήσατε ήδη. Έχω τώρα όμως ένα συγκεκριμένο ερώτημα, παρόλα αυτά. Επεξεργάζεστε ένα σύστημα αναφοράς για αγορές capacity, χωρητικοτήτων. Έχουμε και σχετική πράσινη βίβλο στη Γερμανία και τον προβληματισμό που ακολουθεί διάφορες πραγματογνωμοσύνες που έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο ενέργεια μα, απορρίπτουν αυτέ τις αγορές διότι υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν υψηλότερα, υψηλότερα ε, κόστη συστημάτων και ούτω καθεξής. Και οι εμπειρίες από τις ΗΠΑ δείχνουν επίσης ότι η σωστή διαμόρφωση αυτών των capacity markets είναι και δαπανηρή και χρονοβόρα και χρειάζεται και πάρα πολύ μετά εκ των υστέρων νομοθετική ρύθμιση. Από τη δική σας σκοπιά, πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές, η εισαγωγή αυτών των capacity markets να μην αντιβαίνει στην ίδια την αρχή της ενιαίας αγοράς και να οδηγήσει επομένως σε επανεθνικοποίηση των αγορών ενέργειας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μπούζεκ. Η κυρία Κίρκεν Ντάουλινγκ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Εκφράζω την υποστήριξή μου στα σχόλια του κ. Πέτερσεν για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαχείριση των προτάσεων. Αυτό ο ρόλο θα είναι κρίσιμο. Πάντω, γενικά μου αρέσουν οι προτάσει και ιδίω ο κέριο ρόλο τη αποδοτικότητα τη ενέργεια. Επίση, η πρόθεση που έχετε δώσει στην συνεργασία τη κοινωνία των πολιτών και των πόλεων και ιδίω των Εφιών πόλεων. Μήπως μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο σε ένα σχόλιο που κάνατε απαντώντας στις πρώτες ερωτήσεις για την κοινωνική διάσταση και για τη συνεργασία με την Επίτροπο Τάισεν. Είναι σαφές για μένα ότι ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή θα παίξουν κρίσιμο ρόλο για μια δίκαιη μετάβαση σε αυτή τη νέα ενεργειακή ένωση. Περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν. Τέλος, έχει τονιστεί κατ' επανάληψη ότι πρέπει να συνδέσουμε την Ενεργειακή Ένωση με τη βιομηχανική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το θεματολόγιο της βιομηχανικής πολιτικής είναι και η δέσμευση του διοξιδίου του του άνθρακα. Έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Στην εκλογική μου περιφέρεια, στο ε, βρετανικό T-Side, υπάρχουν εγκατεστημένε βιομηχανίε οι οποίε παίζουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των σχεδίων και που θα οδηγήσουν σε δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχολήσεως και θα διατηρήσουν άλλες χιλιάδες θέσεις απασχολήσεως από τις υπάρχουσες μέσα από αυτή τη διαδικασία ε, αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακος. Η κυρία Καρπαζόν Λούις. Ευχαριστώ. Και εγώ δεν είμαι απόλυτα σύμφωνη. Μάλλον χαίρομαι για τα όσα είπατε για την ανάπτυξη των διαφόρων ε, φορέων ενέργειας και χαίρομαι που μιλήσατε και για την ενεργειακή φτώχεια. Βέβαια δεν μπορούμε να πίνουμε μόνο στα ωραία λόγια, μόνο στα ε, λόγια γενικότερα, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της ενεργειακής φτώχειας. Χρειαζόμαστε και μια γενική στρατηγική που να περάσει σε όλες τις χώρες μέλη. Γιατί οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κατάματα αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να υπάρχουν χώρες που να μαστίζονται από το πρόβλημα αυτό. Χρειάζεται και περισσότερη διαφάνεια ε, για το κόστος της ενέργειας. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη σημαντική αυτή ευκαιρία που διαθέτουμε τώρα. Ας σκεφτούμε το σχέδιο, τον σχεδιασμό Juncker για τις επενδύσεις για να κάνουμε προσπάθεια να λύσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Πρέπει οπωσδήποτε να δραστηριοποιηθούμε. Χρειάζεται ενεργειακή στρατηγική που να είναι άξια του ονόματός της. Thank you, Σας ευχαριστώ, κύριε Μούντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα. Το ένα αφορά τα σχόλια που ήδη έγιναν ε, για την αναγνώριση της σημασίας των κοινοτήτων ε, στην ενεργειακή πολιτική αλλά μιλάτε και για θεσμικούς επενδυτές. Υπάρχουν παραδείγματα στη δική μου την περιφέρεια και σε όλες τις άλλες φαντάζομαι, που είναι συνεταιριστικά τέτοια έργα, αλλά βεβαίως χρειάζονται και κάθε υποστήριξη που μπορούν να λάβουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαν να αποτελέσουν οπωσδήποτε παράδειγμα. Και μετά το άλλο, Υπάρχει αρκετά μεγάλη στήριξη γενικώ και αορίστος, αλλά όταν γίνεται το έργο κοντά μας, βεβαίως ε, τότε δεν υπάρχει η στήριξη και βεβαίως καλό είναι να υπάρχουν κάποια ωφέλη εκεί όπου γίνονται μεγάλα έργα. Και τέλος ε, ανησυχώ για την χρηματοδότηση και το ότι τα παίρνουμε από τη μία τσέπη και τα βάζουμε στην άλλη των φορολογουμένων. Γιατί ακριβώς πρέπει να γίνει μια έρευνα για τις τεχνολογίες, ε, αλλά αν φεύγουν λεφτά από τον προπολογισμό της έρευνας, τα, ουσιαστικά τα παίρνουμε ε, από τις μελλοντικέ ε, τεχνολογίες και ληστεύουμε το μέλλον μας και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ, κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ένα από τα κλειδιά εδώ πέρα είναι να βελτιωθεί η ενεργειακή αυτονομία και να βελτιωθεί η ε, ενεργειακή αυτολισματικότητα, αλλά στο, πλάνο, στο σχέδιο Juncker δεν φαίνονται κάτι τέτοια πράγματα. Αντιθέτω, υπάρχει μείωση σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Πώς συμβάζονται αυτά τα δύο, ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέιρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. com ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα δείχνουν πως η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, ειδικά της αγοράς του ηλεκτρισμού, δεν οδήγησε σε αυτό το οποίο μας λέγατε. Ότι δηλαδή ο τελικός καταναλωτής θα είχε φτηνότερη ενέργεια, αντιθέτως. Οπότε, η ολοκλήρωση από πάνω που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποτέλεσμα βεβαίως στις τιμές παραγωγής και βεβαίως υπέφεραν οι καταναλωτές. Είναι γεγονός αυτό, είναι σαφές. Ε, τούτου λοιπόν ε, δεδομένου η Κομισιόν θα συνεχίσει να μην ε, βλέπει τα προφανή, θα αρχίσει να κάνει κάτι. Βλέπουμε ότι η τιμή του βαρελιού υπόκειται σε διακυμάνσεις που, που με τις ανακοινώσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μελέτη αντικτύπου στο παρελθόν είχε πει ότι θα αντιμετωπίσει, ιδίως με το πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών και την, ε, ε, ανανέωση, τον, την πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να ολοκληρώσουμε, η αγορά του άνθρακα, χαμηλή τιμή του άνθρακα και χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορούν αυτά να συνδυαστούν για την αξιοπιστία του αγοράς άνθρακα που μέχρι τώρα δεν υπήρχε και κυρίως για την ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών. Ε, όλα αυτά δεν πρέπει να συνδυαστούν για να ε, επιτύχουμε για τρόπους επιτυχίας του στόχου μείωσης των εκπομπών ή απλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τρέχει πίσω από τι εξελίξει ε, πίσω ενό μηχανισμού που έχει δείξει στην κοινωνία ότι και αποτελεσματικό είναι και φέρνει στρεπλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λόπες Μπερμαίο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τα λεπτομερή σας ε, σχόλια. Συνήθως δεν έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες, οπότε σας ευχαριστώ. Και ελπίζουμε ότι όλα αυτά που ανακοινώσατε θα υλοποιηθούν. Για το Φεβρουάριο είπατε ότι θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις και θα δείτε αν οι χώρες έχουν ε, υλοποιήσει όσα υποσχέθηκαν. Η Ισπανία έχει καταστρέψει τις ανανεώσιμες πηγές και δεν υπάρχουν ούτε μικροί επενδυτές ούτε μικρές καταναλωτές. Μόνο μεγάλες εταιρείες θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Θα κοιτάξετε να υπάρξει συντονισμός από την ε, οπτική γωνία του ανταγωνισμού για να γίνει κάτι για όλα αυτά. Και φαίνεται ότι κουμάντο κάνουν εδώ οι εταιρείε τελικά. Καθορίζουν τις τιμές και τα πάντα. Ε, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, οι θέσεις εργασίας, όλα αυτά καταστρέφονται σε μεγάλο βαθμό και προκαλούν και ενεργειακή ένδυα. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές, δεν είναι δαπανηρές, δεν ακριβές. Ε, απλώς δεν παίρνουν την ίδια στήριξη με άλλους τομείς. Ε, είμαστε λοιπόν πολύ φιλόδοξοι αλλά πρέπει να τα φροντίσουμε και από την πλευρά της έρευνας και της ε, καινοτομίας. και επίσης ένα αίτημα. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ε, συνδυαστούν στην όλη συζήτηση. Κάτι που μέχρι τώρα δεν φαίνεται να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε, ο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολλά ακούστηκαν ήδη, οπότε θα αναφέρω μόνο αυτά τα οποία θεωρώ σημαντικά. Γνωρίζουμε πως έχετε ένα πολύ περίπλοκο χαρτοφυλάκιο και παρά το ότι ε, είναι δύσκολο να πούμε πως κάποιος επίτροπος έχει πιο δύσκολη δουλειά από κάποιον άλλον, νομίζω πως στην ε, δική σας την περίπτωση είστε επίσκοπος, ε, επίτροπος, με κρίσης. Γιατί η ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο συγκρούσεων, ε, τα έχει δει η Ευρώπη. Και τα βλέπουμε καθημερινά. Αν δείτε δε και τους διάφορους πίνακες δείχνουν πως δεν έχουμε μάθει τίποτα γιατί εξαρτώμεθα βεβαίως από έναν και μόνο προμηθευτή. Και το αναφέρατε βεβαίως ε, και δεν είναι κάτι που θα ήθελα να συστήσω, αλλά θα προτιμούσα να δω λιγότερη φιλοδοξία και περισσότερο ρεαλισμό. Το 2006 είχαμε, ε, μιλούσαμε για το λεγόμενο Ναμπούκο. Μα αν υπήρχε τώρα θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τα δίκτυα καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Και βεβαίως όχι μόνο τις ανανεώσιμες, αλλά να δούμε και τις δικές μας υφιστάμενες ε, πηγές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο πράγματα να λύσει. Το πρώτο είναι η άγνοια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και βιομήχανοι και πολιτικοί ακόμα δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα και την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. Το άλλο ερώτημα είναι πώς ε, θα βρούμε επενδύσεις για τα μακροπρόθεσμα που μας απασχολούν, ανανεώσιμες, όταν βράχει πρόθεσμα δεν μας βοηθάει η κατάσταση. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου και ε, φτηνό πετρέλαιο υπάρχει παντού στην αγορά και υπάρχει κίνδυνος ε, για τις βράχυπρόθεσμες λύσεις. Ποια είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε Μήπως να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Τι απάντηση έχετε να μου δώσετε. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στον κύριο Γκέρεκ. Θα ήθελα και εγώ να πω, κύριε Επίτροπε, πώς 28 οικονομίες σημαίνουν 28 διαφορετικά ενεργειακά μείγματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό εισάγει κοινά συστήματα με βάση το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο, το πρώτο και το δεύτερο, κάτι το οποίο ε, δεν μεταφράζεται σε ίσες ε, ευκαιρίες για όλους, γιατί κάποιες οικονομίες θα χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερο, παραδείγματος χάρη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πώς με βάση την Ενεργειακή Ένωση θέλει να ενισχύσει την αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Παραδείγματος χάρη, η Πολωνία. Εμείς έχουμε άνθρακα. Εάν είναι δηλαδή να έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα μέχρι το 2050, η οικονομία μας θα γίνει η λιγότερο ανταγωνιστική. Είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο. Οπότε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση σημαίνει και καμία νέα ιδέα. Ε, ευχαριστώ. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης είναι οπωσδήποτε η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να αποφευχθούν οι ξαφνικές διακυμάνσεις και να διασφαλίσουμε και σταθερή παροχή ενέργειας. Ένα άλλο θέμα είναι τα έξυπνα δίκτυα, το θέμα της αποκέντρωσης της παραγωγής να έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή και αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης. Αυτή η συνδυασμένη στρατηγική, δηλαδή παραγωγή, μετάδοση, αποθήκευση κοντά στον καταναλωτή, όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί ως θετικά στο παρελθόν και έχει αναγνωριστεί νομίζω ήδη από ανθρώπους οι οποίοι το ζουν. Το ερώτημά μου είναι ποια προσέγγιση υπάρχει από πλευράς Κομισιόν όσον αφορά τον σχεδιασμό των δικτύων για μια ενεργειακή ένωση για να σταματήσουμε ακριβώς αυτόν τον κύκλο της διακύμανσης ε, παροχής ενέργειας και μετά συναντήσατε πρόσφατα τον πρόεδρο ε, του, του δοσού της ε, Gazprom και από την πλευρά της, ε, της εταιρείας δηλαδή δηλώθηκε πως πρέπει να προκαταβάλει το φυσικό αέριο που θα λαμβάνει η Ουκρανία και αυτό σημαίνει λιγότερη ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από ό,τι πληρώνουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μία λύση με μία Ένωση Αερίου. Αλλά πώς συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία σε αυτήν, πώς ακριβώς την οραματίζεστε μια τέτοια Ένωση Αερίου. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Αναμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας κύριε Επίτροπε. Ελίγες προτάσεις ε, για κάθε μέλος τουλάχιστον της Επιτροπής ιτρε. Ευχαριστώ. Ε, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες σας, τις ερωτήσεις σας δείχνουν ε, το ενδιαφέρον που υπάρχει για το κοινό μας έργο. Κυρία Καστίγιο, όταν μίλησα για τα έξυπνα δίκτυα, αυτή ήταν και η ερώτηση της κυρίας ε, Καπέλα, συνειδητοποιούμε πως δεν υπάρχει τρόπος να εισαχθεί έξυπνη ενέργεια στην Ευρώπη χωρίς έξυπνα δίκτυα. Σήμερα μίλησα με τους ε, επικεφαλής της Έντσο ε, Ι, e. ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε για να κάνει ευκολότερη την διασύνδεση των ε, δικτύων ηλεκτρισμού και τους έκανα μία απλή ερώτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το έργο αυτό σε ευρωπαϊκή κλίμακα που θα μα βοηθήσει να έχουμε έξυπνα ολοκληρωμένα δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί γνωρίζω πω στην Ιταλία περιμένουν τα 40 εκατομμύρια έξυπνου μετρητέ. οι Ιταλοί είναι ικανοποιημένοι, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, ε, τα έξυπνα κουτιά και άλλες νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και πρέπει να συνεργαστούμε να δούμε τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσουμε, πώ θα προωθήσουμε την ανάπτυξή της, ε, την διάθεσή της και πώς θα φροντίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνο για τους πλούσιους ε, που θα μπορούν να αποφύγουν τα μέτρα αυτά ή θα μπορούν να αγοράζουν αυτά τα, τα γκατζετάκια. Οι νέοι, οι οποίοι τώρα σπουδάζουν ε, και μπορούν να κάνουν θαύματα με τα smartphone, τα κινητά τους πώς θα αναπτύξουμε την ε, τεχνολογία που υπάρχει και να την έχουν όλοι, φτωχοί, πλούσιοι, όσοι έχουν ψηφιακές ικανότητες, αλλά και άλλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα εφαρμοστούν τα έξυπνα δίκτυα που είναι προϋπόθεση για όλα αυτά τα οποία είπαμε. Μετά μιλήσατε για τη σημασία ενδυνάμωσης των καταναλωτών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ε, βεβαίω οι πολίτες ε, θα μπορούν από το σπίτι τους να αποφασίζουν πότε θα αγοράσουν ηλεκτρισμό. Πρωί, βράδυ, αργότερα, ώρα εχμής ε, και με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Αλλιώς βεβαίως δεν γίνεται τίποτα. Οπότε σαφώς τα έξυπνα δίκτυα είναι πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ε, πώς θα υπάρξει χρηματοδότηση και θα αναπτυχθούν σταδιακά τα έξυπνα δίκτυα. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες ε, αναφέρθηκε στην σημασία της ε, ρυθμιστικής ε, σταθερότητας. Αυτό μου το λένε όλοι οι επιχειρηματίες που συναντώ και είναι πράγματι μια μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει λοιπόν ένας κανονισμός, υπάρχει μια μεταδημοκρατική αλλαγή με μια νέα κυβέρνηση που εξετάζει τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και συχνά υπάρχει η αίσθηση πως ε, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και βέβαια αναρωτιέται κανείς τι σημαίνουν αυτά για τις επενδύσεις, ε, πώς ε, θα επηρεάσει και την εικόνα της χώρας. Ε, δηλαδή αν αλλάζει κανείς νομοθεσία συνεχώς είναι δύσκολο για τους επενδυτές να προγραμματίσουν και εδώ πέρα νομίζω πως μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μεγάλα πλαίσια θα έλεγα και έτσι θα, είναι, θα έχουν την άνεση θα έλεγα οι επενδυτές να επενδύσουν όπου θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν μου λέγατε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή η έννοια της Ενεργειακής Ένωση. θα έλεγα πως είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Κοιτάμε τώρα δηλαδή τις εθνικές λύσεις και αναζητούμε ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη μας να αναζητήσουν λύσεις ε, στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας με την αλλαγή αυτή νοοτροπίας που πρέπει να δούμε μετά τι οικονομία κλίμακας μπορούμε να πετύχουμε, πώς θα αυξήσουμε τις ε, δυνατότητες παραγωγής, ε, να γίνουν καλύτερες οι ανανεώσιμες, τι μπορούμε να κάνουμε με τη βελτίωση του δικτύου LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και το τι θα γίνει και με τους εταίρους μας στην περιοχή και όταν αποδείξουμε πως κάτι τέτοιο δεν συμφέρει μόνο από τη σκοπιά της ενεργειακής ασφάλειας και της αλληλεγγύης αλλά συμφέρει και οικονομικά και επιχειρηματικά νομίζω πως αυτό είναι ένα επιχείρημα καταλητικό για τους Υπουργούς Οικονομικών. Γιατί αν με ρωτήσετε γιατί έχουμε αυτές τις τιμές ε, της ενέργειας, μπορώ να δώσω πολλές απαντήσεις, αλλά ε, η απλή απάντηση είναι τιμή παραγωγής, πόσο κοστίζει η παραγωγή και θα έλεγα πως είμαστε πολύ συγκρίσιμοι στο κόστος παραγωγής με τη ΣΥΠΑ. Αλλά μετά γιατί η διαφορά στην τιμή καταναλωτή. Γιατί υπάρχουν τέλη, φόροι, κόστος δικτύου, και βεβαίως είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν αφορά μόνο την ε, ενέργεια, αφορά τους υπουργού οικονομικών, ε, κοινωνικών ζητημάτων. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η πρόταση φορολογίας ενέργειας, η οποία δεν έχει σημειώσει κάποια πρόοδο. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα τιμολογήσουμε την ενέργεια, τι θα συμπεριλάβουμε, γιατί αφενός παραπονιόμαστε πως είναι ψηλό το ενεργειακό κόστος, απ' την άλλη δεν θέλουμε να δούμε τι άλλα στοιχεία ε, μπορούμε να ενσωματώσουμε στην ε, τιμή καταναλωτή και θέλουμε οι πολίτες, οι καταναλωτές ε, να τα πληρώσουν. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η δομή της τιμής ενέργειας και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ένας άλλος βολιστής ρώτησε για την ασφάλεια προμήθειας και τη λεγόμενη λύση Turk Stream. Τα συζητήσαμε αυτά με τον κύριο Αλεξέη Μίλερ για τη μία νέα προσέγγιση. Κοιτάξτε, εγώ απορώ λίγο, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζονται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, αλλά τόσα είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη 15 ε, και 15, 30 δηλαδή χοντρικά το σύνολο και θέλουμε να φύγουμε από τη διαδρομή της Ουκρανίας ε, και να πάμε στην Τουρκία. Και υπάρχουν ε, όμως άλλα 33 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που περισσεύουν. Τι θα τα κάνουμε αυτά, δεν υπάρχουν υποδομές. Και δεν νομίζω πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες απλά θα αλλάξουν τα συμβόλαια και θα πούνε πως ε, θα τα πάρουμε όλα τώρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα αλλάζει απλά ο τόπος παράδοσης. Πρέπει να το ξαναδούμε λοιπόν αυτό και δεν έχω δει μέχρι σήμερα καμία οικονομική βιωσιμότητα για να κλείσει η διαδρομή της Ουκρανίας. Δεν είναι λοιπόν οικονομική η απόφαση, είναι πολιτική και ελπίζω πως ε, θα μπορούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και να δούμε αυτή την πρόταση από οικονομική σκοπιά γιατί η υποδομή υπάρχει, είναι ανεπτυγμένη βεβαίως είναι σαφές πως πρέπει να γίνουν τεράστιες μεταρρυθμίσεις στο ουκρανικό σύστημα μετάδοσης αερίου, αλλά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να αναβαθμίσουν το σύστημα, να υπάρξει κάποια διαφάνεια, αλλά είναι πολύ σημαντική η διαδρομή αυτή για την Ουκρανία, κεντρική και ανατολική Ευρώπη ε, και νομίζω πως είναι και πάρα πολύ σημαντικοί πελάτες της Ρωσίας. Οπότε Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάτι πιο λογικό, αλλά δεν θα περιμένουμε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε ενδεχόμενο. Θα επεξεργαστούμε ένα νέο σχέδιο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, τη βελτιστοποίηση των υποδομών LNG, έτσι ώστε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι από ό,τι στο παρελθόν και βεβαίως ε, μέρος αυτού αποτελεί και η συνεργασία μαζί σας για την επανεξέταση της ασφάλειας ε, παροχής ε, φυσικού αερίου και θέλουμε να μάθουμε ε, και από τις τελευταίες οδηγίες. Και είμαστε νομίζω πολύ πιο προετοιμασμένοι για τυχόν μελλοντικά προβλήματα. Κύριε Ντάλα ανέφερε το το φυσικό αέριο της Μεσογείου τι θα κάνουμε, μα συμβαίνει ήδη αυτό. Στη Ρώμη αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τρεις πλατφόρμες για την Μεσόγειο, για, τον, για ηλεκτρισμό, για αέριο και ανανεώσιμες. Και ήδη αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις ε, ειδικών για το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες ε, περαιτέρω προμηθειών από τη Βόρεια Αφρική, αλλά επίσης συζητάμε και με τους Κύπριους ε, και Ισραηλινούς εταίρους μας ε, το τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδέσουμε ακριβώς ε, τα νέα αυτά κοιτάσματα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αερίου. Μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Νομίζω πως η Μεσόγειος θα γίνει πάρα πολύ σημαντική ως προμηθευτής αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκέρεκ ανέφερε το ότι δεν είναι ολοκληρωμένη η εσωτερική αγορά και συμφωνώ οπωσδήποτε μαζί σας. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Λογισμικό οπωσδήποτε και υλικό που πρέπει να αναβαθμιστεί. Εγώ λογισμικό θα έλεγα όλα αυτά τα τα διοικητικά εμπόδια, φραγμούς που απλά δημιουργούν εμπόδια για το εμπόριο ενέργειας που πραγματικά καθίσταται αδύνατον. Έχω δει τη χαρτούρα δηλαδή, είναι οι φάκελοι τεράστιοι. Και πρέπει να εναρμονίσουμε τους κωδικούς των δικτύων να μιλάνε μεταξύ τους οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρισμού, να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορεί να ρεύσει η ενέργεια. Και χρειάζονται ακριβώς ε, διασυνδέσεις με το υλικό, τις δυνατότητες δηλαδή, να υπάρχουν δυνατότητες να στείλουμε την ενέργεια στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτό το έργο κοινού ενδιαφέροντος που νομίζω χρειάζεται, όπως είπα, πολύ στενότερη παρακολούθηση για να είμαστε σίγουροι ότι εργαζόμαστε σε έργα τα οποία είναι βιώσιμα και αφορούν ακριβώς την ρευστότητα, θα έλεγα, της αγοράς ενέργειας και θα καταστήσουν πραγματικότητα την εσωτερική αυτή αγορά. Η κυρία Καλάς μίλησε για το Acer και τους άλλους φορείς που δημιουργήθηκαν ε, από ρυθμιστικούς φορείς ή διαχειριστές ε, δικτύων και ειλικρινά έχω μεγαλύτερες προσδοκίες από όλους αυτούς γιατί οι ευρωπαϊκοί αυτοί φορείς πρέπει να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε πρακτικές λύσεις ε, για το πώς θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Νομίζω πως ε, βεβαίως ε, πάντα βοηθάει το να έχουμε τις συμβουλές των ανθρώπων που δουλεύουν κάθε μέρα πάνω στο αντικείμενο. Αλλά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Μην κοιτάμε το πρόβλημα της ενέργειας μόνο εντός των συνόρων μας, αλλά να αναζητήσουμε λύσεις πανευρωπαϊκές. Έχει σημειωθεί νομίζω αρκετή πρόοδος ήδη, τα είδαμε και το πρωί με τον κύριο από την Έντσο ή που μου είπε πως ε, βεβαίως αναμένει πολύ καλύτερη αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη για να υπάρχουν λύσεις ε, στην Ευρώπη και όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων. Η κυρία Μπερές ε, αναφέρθηκε στην τιμή του άνθρακα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι Νομίζω πως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν σε ένα αποθεματικό σταθερότητα της αγοράς, τα ανοιχτά ζητήματα, τι θα κάνουμε με τις 900 ε, εκατομμύρια σε άδειε που έχουν μείνει μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα ψυγείο θα έλεγα εντός αγωγικών και να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε αργότερα να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην έρευνα και ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα γι' αυτό, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτή θα ήταν μια δυνατότητα και βεβαίως μετά αντιλαμβάνομαι πως ε, υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα κάνουμε με το θέμα της διαρροής άνθρακα και θα το συζητήσουμε και με την Επιτροπή Ένβη, αλλά μπορούμε νομίζω στα εκτιμώντας να κάνουμε μία δήλωση της ε, Κομισιόν που θα λέει πως θα πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό ε, και να συμπεριλάβουμε όλους τους ενδιαφερόμενους γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στο θέμα της ε, σταθερότητας της αγοράς γιατί έτσι θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και για την τιμή του άνθρακα. Θα δείξουμε στους ε, επιχειρηματίες πως ε, σοβαρολογούμε και πως υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για μετά το 2020 για να δούμε πως θα προγραμματίζουν τις επενδύσεις γιατί γνωρίζετε πως η διαδικασία διοδότησης είναι πάρα πολύ δύσκολη χρειάζεται 10 χρόνια για να προγραμματιστεί ένα έργο και βεβαίως η δουλειά που γίνεται τώρα νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει. Δεν μιλάω για την διάσκεψη των Παρισίων, όπου θέλουμε... Θέμε να πάμε πραγματικά με πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα έχουμε να επιδείξουμε όσο θετικά. Μετά αυτό το οποίο αναφέρθηκε την κυρία Ντάλιν για τον κοινωνικό διάλογο, οπωσδήποτε μας απασχολεί ε, και με την κυρία Τάισεν ε, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε να συμπεριλάβουμε την ενέργεια στον κοινωνικό διάλογο. Ε, τα έχουμε συζητήσει με την Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για μια just transition, όπως λέμε, μια δίκαιη μετάβαση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κόσμο που δουλεύει στον τομέα, ε, που πρέπει πιθανώς να αναβαθμιστούν οι δεξιότητές τους. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν θύματα στην αγορά εργασίας λόγω της ενεργειακής αυτής μετάβασης και πρέπει να το συζητήσουμε με τους ε, κοινωνικούς εταίρους πώς θα το αποτρέψουμε αυτό και κοιτάμε τώρα τις λεπτομέρειες πώς θα οργανωθεί ο κοινωνικός διάλογος. Πώς θα χρηματοδοτηθεί λοιπόν η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η σχετική έρευνα. Ε, νομίζω πως έχουμε κάποια καλά προηγούμενα εδώ πέρα. Τώρα έχουμε το νέο ταμείο των 400 το λεγόμενο και νομίζω πως θα στείλουμε το μήνυμα στις ιδιωτικές εταιρείες ε, να εμπλακούν και θα βλέπουν πλέον πως θα συμφέρει και οικονομικά κάτι τέτοιο γιατί ε, το ίδιο ισχύει βεβαίως και για κάποια ζητήματα άνθρακα, καθαρού άνθρακα κτλ. Και πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και ότι χρησιμοποιείται βεβαίως σε βιομηχανική κλίμακα. Ευχαριστώ τον κυρία Μούντι που τόνισε την σημασία της εμπλοκής των κοινοτήτων, συνεταιρισμών, στις συζητήσεις αυτές, γιατί κάθε σύστημα διαφέρει ελαφρώς. Άκουσα πάρα πολλά θετικά πράγματα για τα πράσινα ε, ταμεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βοήθησαν πάρα πολλούς δήμους να αυξήσουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα σπιτιών, διαμερισμάτων και βεβαίως ε, χρειάζεται ευελιξία για την κάθε χώρα γιατί γνωρίζω πως το σύστημα και οι νόμοι ε, συχνά διαφέρουν, ε, οι αρμοδιότητες των Δήμων διαφέρουν, αλλά τέλος πάντων πρέπει γενικά να υπάρχει το σκεπτικό πως είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και να βρούμε μία λύση και να το παρουσιάσουμε αυτό ως παράδειγμα, όχι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και επιχειρηματικό. Πολλοί από εσάς αναφερθήκατε στις ανανεώσιμες ξεχνάμε λίγο πως ε, υπάρχουν νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ανανεώσιμες που αντικατοπτρίζουν θα έλεγα την ε, οριμότητα των τεχνολογιών αυτών που υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη και τώρα τι γίνεται. Περνάμε από εγγυημένε τιμές ε, σε πριμ δηλαδή τα τέλη που είναι πάνω από την κανονική τιμή αγοράς, ε, προ ένα σύστημα δημοπρασιών μέχρι το 2017 για να ενσωματωθούν πλήρως οι ανανεώσιμες πλέον στην αγορά ενέργειας, στον ανταγωνισμό με τις άλλες πηγές ενέργειας γιατί θεωρούμε πως η ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών πλέον γίνεται πιο φτηνή και θα είναι πιο ανταγωνιστική και θα βοηθήσουμε να υπάρξει περισσότερος ε, ανταγωνισμός στην αγορά και καλύτερες τιμές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ε, για τον κύριο Τοσενόφσκι μία απάντηση. Αν πάει κανείς σε διεθνείς διασκέψεις τώρα υπάρχει ένα νέο θέμα. Η νέα γεωπολιτική της ενέργειας, κάτι το οποίο ακούμε συνέχεια λόγω της κατάστασης με το πετρέλαιο και τις επιπτώσεις που έχει σε κάποιες χώρες ε, όπου βλέπετε ήδη ταραχές λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης ε, μέχρι τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, της σχέσης με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε σαφείς για τις προτεραιότητές μας ε, τις δυνατότητες διαφοροποίησης, ο νότιος διάδρομος και είμαστε έτοιμοι να το χρηματοδοτήσουμε. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, τους εταίρους μας, να μην δημιουργήσουμε νέα εμπόδια, αλλά να ανοίξουμε το δρόμο και να διδαχτούμε από το παρελθόν. Και τέλος, τελευταία παρέμβαση του κυρίου Έριξεν αναφερόμαστε στις ανανεώσιμες και στο ότι δεν χρειάζονται μόνο έξυπνα δίκτυα αλλά και αποθήκευση της ενέργειας. Αν ξαναδείτε λοιπόν τις διαφάνειες και το που βρισκόμαστε στην έρευνα και την ανάπτυξη θα δείτε πως δυστυχώς όταν μιλάμε για αποθήκευση είμαστε πίσω από τους Ασιάτες ανταγωνιστές μας. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος έτσι ώστε όχι μόνο να παράγουμε αλλά και να μεταφέρουμε και να αποθηκεύουμε ανανεώσιμη ενέργεια και έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Γκέρεκ για ενέργεια και τα λοιπά. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω τουλάχιστον σε όλους τους ομιλητές, να δώσω μία απάντηση στον καθένα και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και αναμένω τη μελλοντική μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον για όλους μας. Περάσαμε πάνω από δύο ώρες μαζί. Σχεδόν νέα περάσατε κύριε Επίτροπε, όπως πριν από ένα τρίμηνο. Λίγο, λίγο λιγότερο. Τέλος πάντων, οριακά ε, λιγότερο. Απλώς να πω και τη δική μου τη γνώμη. Η υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας είναι το πλέον σημαντικό για το εγγύς μέλλον, διότι ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες και ο στόχο δεν είναι να πάνε τα κράτη-μέλη στο ΔΕΚ. Ε, αυτό έτσι κι μπορεί να γίνει, αλλά καλύτερο είναι να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναζητηθούν ε, εναλλακτικέ λύσει. Και αναμένουμε τι επόμενε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δικού χάρτε για την Ενεργειακή Ένωση, για, τα, για το Παρίσι, για του διασυνδέτε. Πώ τα προβλήματα αυτά μπορεί να ε, αντιμετωπιστούν από κοινού. Είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας και σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για πάνω από δύο ώρες. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Μπούζεκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε και άλλο ε, επίση σημαντικό θέμα στην ημερησία διάταξή μα. Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις, αλλά Ο πρόεδρος Μπούζεκ. Κυρίες και κύριοι, α έρθουμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσια διάταξή μας, το οποίο είναι, σας παρακαλώ, κτυπ κτυπ η σφύρα. Παρακαλώ κύριε και κύριοι, καθίστε κάτω. Αν δεν επιθυμείτε να παραμείνετε στην αίθουσα, εγώ θα λυπηθώ πολύ, δεν μου φαίνεται καλή ιδέα, αλλά μπορείτε να αποχωρήσετε. Εάν όμως αποχωρήσετε, παρακαλώ ήσυχα. Ευχαριστώ. Τώρα το άνοιγμα της ανάπτυξης μέσω της γαλάζιας οικονομίας που είναι το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας για σήμερα το απόγευμα. Και αν με επιτρέπετε να ζητήσω πρώτα από τον εισηγητή μας κύριο Φερέιρα να αναπτύξει το θέμα του. Έχετε το λόγο αγαπητέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα την πρόθεση σήμερα εδώ να περάσω σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μόνο αυτό. Ήθελα μια γενική και προκαταρκτική ανταλλαγή για το ποια θα είναι η προσέγγιση μας για την έκθεση αυτή, τους στόχους της και το τοπίο στο οποίο θα κινηθεί. Πάντως μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις ε, προκαταρκτικές αντιδράσεις και των ε, σκιωδών συγητών, των συναδέλφων και όσων εκπολείπων ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, αλλά και όσων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τους απασχολεί. Ξέρουμε ότι οι θάλασσες, οι ωκεανοί είναι ανέκαθεν πηγή πόρων για την ανθρωπότητα η σχέση μας με τους θάλασσες και τους ωκεανούς πλήγει ιδίω στο τελευταίο ε, μισό του 20ου αιώνα, ιδίω τα τελευταία 50 χρόνια και υπήρξε μια σοβαρή ποιοτική αλλαγή. Οι παραδοσιακές ε, ανάρχες δραστηριότητες όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η αλληλεία και άλλες δραστηριότητες αντικαθίστανται από νέες δραστηριότητες, αναδυόμενες, εάν μπορώ να το πω έτσι, που σκοπό έχουν να εξερευνήσουν τους ανεξάντλητους πόρους των θαλασσών και των ωκεανών να, ε, ή έστω να ε, εξερευνήσουν με άλλο τρόπο αυτές που ήδη ήταν γνωστές. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ποιοτικέ αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Από τη μια έχουμε την μείωση της σημασίας των θελάσσιων μεταφορών, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα, επόμενα χρόνια ωστόσο, έχουμε σημαντική αύξηση των ε, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις θάλασσες και τον ωκεανό, όπως ο τουρισμός, ο ναυτικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός αλλά και αυξανόμενη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ε, ενεργειακών πόρων των ωκεανών, ιδίως ε, των ορυκτών, ε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όπως έχουμε διαπιστώσει ότι εκτός από τις χρυσές πηγές υπάρχουν και θαλάσσιες. Και πέραν των μελετών και του ενδιαφέροντος εξερεύνησης ε, των ε, πόρων αυτών των θαλασσών υπάρχει και η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού στα κύματα, τα ρεύματα, την παλήρια, την ε, θαλάσσια βιομάζα για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, ε, έχουμε βιολογικές ε, τεχνολογίες που σχετίζονται με την θάλασσα. Ε, εν τέλει, όλη αυτή η αλλαγή μας φέρνει αντιμέτωπους σήμερα με μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Η απόκριση που θα δώσουμε σε αυτές τις προκλήσεις εξαρτάται από την καλύτερη γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τους τεράστιους πόρους των θαλασσών μας, των ωκεανών μας, των παράκτιων ζωνών. Πολύ συνοπτικά θα έλεγα ότι υπάρχουν παραδοσιακοί τομείς που συνδυάζονται με αναδυόμενους, όπως η αλληλεία, οι θαλάσσιες, ε, οι ποτάμιες μεταφορές, ο τουρισμός, η ναυπηγική και η ναυτική τέχνη, όλα όσα έχουν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές και την αλλαγή του τοπίου στις παράκτης ζώνες. Αυτά είναι τα παραδοσιακά στοιχεία και έχουμε και νέους τομείς όπως η ε, ενεργειακή πόρη, η ορυκτή πόρη, η βιολογική τεχνολογία, η πολιτιστική διάσταση με πολλές προκλήσεις. Σε όλους αυτούς τους τομείς διαμορφώνεται ένα πλαίσιο για την έκθεσή μας που έχει να κάνει με την καινοτομία της γαλάζιας οικονομίας. Το ερώτημα είναι αν θα επικεντρωθούμε μόνο στους αναδυόμενους τομείς ή αν πρέπει να δούμε την καινοτομία και από την ευρύτερη πρόπτικη που καλύπτει και τους λεγόμενους παραδοσιακούς τομείς. Αρκεί να θυμηθούμε ότι η αλληλευτική δραστηριότητα και αυτή της ηχθοκαλλιέργειας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις ως προς την βιωσιμότητα, την επιλογή των μεθόδων, την καταπολέμηση της ε, παράνομης και λαθρέας αλίας, Όλα αυτά μπορεί να περνούν από την καινοτομία που έχει ένα τεράστιο δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση όπω ε, έχει αναφερθεί. Ε, η ίδια η δατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει προκλήσει ω προ την αποτελεσματικότητα τη παραγωγή, των αυτόχθονων ε, ειδών, των θαλάσσιων και ποτάμιων ε, μεταφορών είτε κατάντη είτε ανάντη της ε, ναυπηγικής ενό τομέα όπου η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια γνώρισε αρνητικές εξελίξεις επειδή απελευθερώθηκαν οι αγορές και άνοιξαν οι ασιατικές αγορές ναυπήγησης ε, αυτή η αρνητική εξέλιξη μπορεί όμως να αναχαιτιστεί αποτελεσματικά εφόσον επικεντρωθούμε στην καινοτομία και την ιδιαίτερη εξειδίκευση, ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία και καταπολέμηση του ανταγωνισμού των αγορών της από Αυτό δείχνει ότι οι τομείς αυτοί έχουν μέλλον μπροστά τους. Ήδη ανέφερα τις ε, θαλάσσιες περιοχές και την προστασία των παράκτιων ζωνών Κάτι που και πάλι μπορεί να συσχετιστεί με τον τομέα της καινοτομίας, αλλά και με άλλους αναδυόμενους τομείς, την ε, ε, εξερεύνηση των ορυκτών πόρων, των ενεργειακών πόρων, τη χρήση των βιολογικών τεχνολογιών, και εδώ πάλι είναι εμφανή η σημασία της καινοτομία και ο ρόλος της στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παραγωγή ανάπτυξης πλούτου και οικονομικής πρόοδου. Μερικές παρατηρήσεις για να ολοκληρώσω αυτές τις παρατηρήσεις που είναι τόσο συνοπτικές ήθελα να τις ακούσετε ως μέρημνες που κατά κάποιο τρόπο καλό θα ήταν να αναφερθούν στην έκθεση. Σε πρώτη φάση αφορούν την ε, ευαίσθητη ισορροπία των πόρων που συζητούμε, που με την αξία τους, την ε, ποικιλία τους, τις περιβαλλοντικές και οικολογικές λειτουργίες τους απαιτούν να προστατευθούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό ε, φέρνει σε προκατονιστικό ρόλο τα κράτη για την προστασία των συγκεκριμένων πόρων, ώστε να προστατευτεί πάνω από όλα το κοινό, το δημόσιο συμφέρον. Υπέρ των, ε, μάλλον ε, περισσότερο από ό,τι τα τομεακά ή εταιρικά συμφέροντα. Επίσης, ναι, ναι κατάλαβα ότι εξελίγει το χρόνο, θα ολοκληρώσω. Απλώς, πέραν κάποιων ε, σημείων που είχα ετοιμάσει, Υπάρχουν και θέματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο των διαφόρων δομών που παρεμβαίνουν σε αυτό το τομέα και να δούμε και οι δομές και τα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως με το πρόγραμμα πλαίσιο και άλλα, κατά πόσον είναι ε, επαρκή και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του τομέα αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Θα έχετε και άλλη ευκαιρία να πάρετε το λόγο στο τέλος της συζήτησής μας. Οι σκιώδεις εισηγητές μας τώρα. Η κυρία Νταλή. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα για αυτή τη λεπτομερή παρουσίαση. Όταν άρχισα να μελετώ τον τοσχέ αυτό, άρχισα να κάνω κάποιες έρευνες και είδα να παράθεμα της Επιτρόπου Γκίνγκεν Γεώργιεν, η οποία είπε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τον βυθό της θάλασσας και τις κινήσεις της σελήνης. Για σκεφτείτε το αυτό σε σχέση με τη γαλάζια οικονομία και τους ωκεανούς με τις θάλασσες που μας περιβάλλουν λέει ότι η γαλάζια οικονομία μπορεί να παίξει ένα ρόλο και στην επιστηστική ασφάλεια ακόμα σε τέτοια θέματα. Η, η καινοτομία και η γαλάζια οικονομία μπορεί να μας ε, βοηθήσουν στους σκοπούς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ε, Ιδίω σε καιρό που μιλάμε τόσο πολύ για κρίση. Ήθελα λοιπόν πρωτίστως να ευχαριστήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα δράση για την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αναφέρομαι στου τομεί που και ο κ. Φερέιρα ε, ανέφερε, αλλά και άλλου, όπω η δατοκαλλιέργεια, η θαλάσσια η παράκτια, και ο παράκτιο τουρισμό, οι γαλάζιε τεχνολογίε, η γαλάζια ε, διαχείριση των ωκεανών εδώ έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στη θαλάσσια και ναυτική οικονομία. Γιατί μπορούμε ε, με νέες τεχνολογικές λύσεις και offshore να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά και με τον γαλάζιο τεχνολογικό τομέα. Επίσης, πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε να πετύχουμε το εξής, να αποκτήσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται, με εξειδικευμένη εκπαίδευση. Αυτή νομίζω είναι η ευκαιρία μας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μακροπρόθεσμα για να έχουμε περισσότερη έρευνα και όλος ιδιαίτερος έρευνα σε επίπεδο συνεργασιακών σχέσεων. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να έχουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς την κοινοτομία όπου θα προωθηθούν μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων αλλά και σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα σε αυτόν τον χώρο. Τρία σημεία λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρω το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας με ε, εξειδικευμένου και καταρτισμένους επαγγελματίες, αλλά και με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων για εργαλεία και εξοπλισμούς. Έπειτα, νομίζω ότι όλα τα κατημέλη έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαρματίσουν εδώ, όμως θα ήθελα περισσότερες κοινέ δράσεις, ιδίως επειδή πολλά σημαντικά θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Εδώ αναφέρομαι σε τρεις συγκεκριμένους τομείς, να καλυφθούν οι ελλείψεις ε, των γνώσεων ε, για τις ευρωπαϊκές θάλασσες και τους ωκεανούς, να συντονιστούν οι προσπάθειες μελέτης και επιστήμονες ε, καθώς και οι επαγγελματίες με δεξιότητες να, εργαστούν, να συνεργαστούν σωστά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και ο ιδιωτικός τομέας έχει τον ρόλο διαδραματίσει. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να εντοπίσει και να διαρθρώσει ανάγκες για έρευνα στην αγορά και να ε, προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα. Για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι η καινοτομία στην γαλάζια οικονομία μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακάμψει, να βοηθήσει τι παράκτητε περιοχέ να αναπτυχθούν και οι σχετικές δράσεις της πρότασης έχουν τεράστιο δυναμικό για να βελτιώσουν τους ωκεάνιους πόρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να, να δημιουργήσουν απασχόληση και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και για όλους αυτούς τους σκοπούς ε, ανυπομονώ για τη συνεργασία με τους συναδέλφους στην Επιτροπή αλλά και τον κύριο Φερέρα και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε από κοινού να απαντήσουμε τις ερωτήσεις του για το ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας ε, καθώς προχωρούμε στην ε, σύνταξη της έκθεσης Πρόεδρος, ευχαριστούμε ε, για την τοποθέτησή σας εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και τώρα ο συνάδελφος Μαραγκάλα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως εξήγησε ήδη ο φίλος Φερέιρα, ανοίγεται μια θαυμάσια ευκαιρία για να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Γιατί κάπως το θέμα έχει αμεληθεί από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ναι μεν έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Το έγγραφο εργασίας είναι καλό. Η εντύπωση που έχω είναι ότι πρέπει να ρηχτεί φως στο έργο αυτό και με πλήρη συνεργασία. Πρέπει να είναι πιο στοχευμένο το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να βασίζεται σε ένα σχέδιο για την εκμετάλλευση των θαλασσών με ανάπτυξη και με ορθή χρήση των πόρων των ωκεανών. Όπως είπε ο κύριος Φερέιρα, πρέπει να βάλουμε κάπου μια κόκκινη γραμμή. Πρέπει να είναι η προστασία δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι πρέπει να οριοθετείται η οικονομική εκμετάλλευση των θάλασσών. Πρέπει δηλαδή να προστατεύεται το περιβάλλον και να προστατεύεται το δημόσιο όφελος. Ο κίνδυνος με το έγγραφο εργασίας είναι ότι θα προωθήσει υπερβολικά την εκμετάλλευση των θάλασσων. Πρέπει να το εξισορροπήσουμε προωθώντας και άλλα προγράμματα για την προστασία άλλων συμφερόντων. Βεβαίως συμφωνούμε με την αξίωση για περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη έρευνα, πράγματα που είναι απαραίτητα για να προχωρήσουμε. Ορισμένες από τις αυτές είναι υπερβολικά ευρέως ορισμένες. Χρειάζεται λοιπόν πιο συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να είναι και δυνατόν να ελεγχθούν και να μετρηθούν οι επιπτώσεις τους δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση των βιοτόπων για να γνωρίζουμε και ποιον πλούτο κρύβει η θάλασσα. Τώρα για τις παράκτητες περιοχές νομίζω ότι κάθε καινούρια γνώση που κατακτούμε θα πρέπει να μας οδηγεί και στην ανάληψη μιας προσπάθειας για την προστασία των ειδών, προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πέρα από τα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτων που αναφέρονται μέσα στο κείμενο, χρειάζεται μια ξεκάθαρη στρατηγική με σαφείς στόχους και σαφείς δείκτες και η στρατηγική αυτή βέβαια πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της γαλάζιας ανάπτυξης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Άλλος κανείς? Εσείς κύριε μου. Ναι, ευχαριστώ. Σύντομα. Για το θέμα των ε, θέσεων εργασίας. Εγώ εκπροσωπώ την Νότια Ανατολική Αγγλία που έχει και πολύ μεγάλη ακτογραμμή αν έχετε κοιτάξει το χάρτη. Και σε αυτή την ακτογραμμή υπάρχουν πολλές στερημένες κοινότητες όπου πολλοί εκεί δουλεύουν σε αβέβαιες θέσεις εργασίας και με χαμηλούς μισθούς. Αν λοιπόν η γαλάζια οικονομία μπορέσει να προσφέρει καλές δουλειές, είναι σημαντικό αυτό. Καλής ποιότητας δουλειές με κάποια μακροπρόθεσμη προοπτική, ιδίως για κοινότητε και περιοχές που τις χρειάζονται απαραίτητα. Ορίστε εσεί. Α, καλά, έχω εγώ τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, τον κύριο Κίνγκ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται πράγματι για σημαντικό μέρος της δουλειάς της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και οι δουλειές που μπορούν να προέλθουν από τη γαλάζια οικονομία είναι σημαντικά και ότι μπορούν πράγματι να αυξηθούν κι άλλο. Με την έννοια αυτή είναι καλά τα νέα, πώς δηλαδή μπορεί να συμβάλλει η γαλάζια οικονομία στο να ξαναβρει ο κόσμος δουλειά σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως βέβαια σε παράκτιες περιοχές. Το 2012 εκδώσαμε ανακοίνωση που εξέταζε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της γαλάζιας οικονομίας και υπολογίζαμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 2 με 3 εκατομμύρια παραπάνω θέσεις δουλειάς μέχρι το 2020, αν ληφθούν βέβαια τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής. Ίσως αυτό να σας φανεί υπερφιλόδοξο, Έχουμε εξετάσει όμως με περισσότερη λεπτομέρεια διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα τον ε, τομέα της ωκεάνιας ενέργειας. Έχουμε κάνει και ένα Energy Forum για να ε, συνέλθουν εκεί να ασχοληθούν, να συζητήσουν μάλλον όλοι αυτοί που ασχολούνται με την ενέργεια των κυμάτων, με την ενέργεια της παλήριας κλπ. για να αναπτυχθεί μια πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να δώσει πολλές δουλειές πολλές θέσεις εργασίας και που να είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλή σε εκπομπές καυσαέριων. Το ζήτημα εδώ είναι δεξιότητες και καινοτομία. Η γαλάζια οικονομία δεν θα μπορέσει να αποδειχθεί επιτυχής αν δεν υπάρχει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η δε έρευνα που θα χρηματοδοτήσουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και οι χώρε μέλη πρέπει να συμβάλλουν ή θα μπορέσουν να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη άλλων τομέων και όχι μόνο των νεοφιών αυτών τομέων όπως εξόριξη ορυκτών από το βυθμένα της θάλασσας και άλλα σχετικά, αλλά και οι παραδοσιακές βιομηχανίες όπως αλία και ναυπηγική. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 προβλέπει συγκεκριμένα κονδύλια για την γαλάζια οικονομία και έναν αριθμό έργων, ένας αριθμός έργων μάλλον, έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα προώθησης 2014-2015. Αλλά αυτή η καινοτομία δεν μπορεί να προέλθει από το κενό. Η καινοτομία της γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να προκύψει από μια συνεργασία των ερευνητών με την βιομηχανία, του ερευνητικού εργαστηρίου με την ε, βιομηχανία. Διότι εκεί βρίσκεται το κλειδί για να προκύψουν οι δουλειές η πλατφόρμα έρευνας που προτείνουμε με την ανακοίνωσή μας ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ρίξει φως στις προόδους που έχουν γίνει από τους ερευνητές μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και ελπίζουμε ότι και το φόρουμ Business και το οποίο ε, έχει ε, διοργανωθεί θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια αποκατάσταση ενός συνδέσμου μεταξύ φορέων καινοτομία και βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας που μας εξηγήσατε τη θέση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποιον λόγο δηλαδή προωθεί αυτές τις δραστηριότητες. Τώρα κύριε Σιγητά, εσείς αγαπητέ Περέιρα, κάντε την τελική σα ε, σύνοψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σημείωσα προσεκτικά τις απόψεις που εξέφρασαν εδώ οι συνάδελφοι και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Υπάρχει αυτή μεγάλη ανησυχία για το δυναμικό ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλος ο προβληματισμός για θέματα που δεν ανέφερα στην αρχική παρέμβαση, για την ε, γρήγορο, για το γρήγορο σχηματισμό μιας εργατικής δύναμης, ενός ανθρώπινα δυναμικού με σκοπό την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να το δούμε και μέσω της έκθεσης και μέσω των εξελίξεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια και το κατά πόσον υπήρξε απεπένδυση από τα υψηλά προσόντα ή της, την υψηλή εξειδίκευση ε, στον χώρο των θαλάσσιων ε, θέσεων εργασίας πρέπει να σχετίσουμε τους στόχους του προγράμματος με τους στόχους της έρευνας όπως αναφέρθηκε και το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζοντας 2020 Ήδη έχουν ε, προεπιλεγεί κάποια προγράμματα σε αυτόν τον τομέα, οπότε πρέπει να γίνει μια προκαταρκτική αξιολόγηση, αναγκαστικά ιδιαίτερα προκαταρκτική στη φάση που βρισκόμαστε, αλλά για να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα πλαίσιο της έρευνας, ε, λαμβάνοντα υπόψη και τις πρόσφατες περικοπές στο πρόγραμμα αυτό. Να δούμε μήπως πρέπει να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των περικοπών στο πρόγραμμα πλαίσιο σε το συγκεκριμένο χώρο. Με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ προς την βιωσιμότητα, ναι, είναι μια μέρημνα που θα απασχολήσει όλους το, τα κεφάλαια της έκθεσης. Είναι μια ε, να μην επαναλάβουμε στη θάλασσα όσο κάναμε στραβά στην ξηρά. Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η πρόπτικη πρότυπα αξιοποίηση των πόρων που αποδείχθηκαν επιβλαβή να μην προταθούν και για τη θάλασσα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και έπειτα υπάρχει και η συνολική πρόπτικη της έκθεσης να μην επικεντρωθούμε στον ένα τον άλλο τομέα, στον άλλο αναδυόμενο τομέα, στους θαλάσσιους πόρους, αλλά να έχουμε μια συνολική θεώρηση. Το είπαν οι συνάδελφοι, το είπε και ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεθνή ΜΑΡΕ. Και συμφωνώ απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω περισσότερες, περισσότερα σχόλια. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία σε μελλοντικέ συνεδριάσεις να συζητήσουμε το τόσο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Ένα θέμα που θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον και επειδή τα είδαμε και με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα το συζητήσω καλύτερα και με τους συναδέλφους. Καλό θα ήταν να οργανώσουμε μια κρόαση στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό, Δυστυχώ όμω το πρόγραμμα για την ώρα είναι πολύ αυστηρό, πολύ σφιχτό, δεν έχουμε πολύ περιθώριο. Μόλι όμω βρεθεί η ευκαιρία θα πρέπει να δούμε μήπω μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τη συμμετοχή άλλων φορέων στην εκπόνηση τη έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Την πρόταση αυτή τη στέλνουν οι συντονιστέ και θα την σκεφτούμε την πρότασή σας. Ε, η έκθεση θα εξεταστεί 24 και 25 Μαρτίου και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 21 Μαρτίου. Αυτά για σήμερα και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας 23 Φεβρουαρίου. 3 με 6.30 και 24 Φεβρουαρίου 9 με 12.30. Και 3 με 6.30. 23 και 24 Φεβρουαρίου λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε τρεις εβδομάδες.